Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη προβλέπεται κοινή συζήτηση όσον αφορά την πολιτική συνοχή σε Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκθεση Κοτσολίνο για την αστική αναβάθμιση ως συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επίσης την έκθεση Βόγκαν, ρόλος της εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή έκθεση Κολάρσκα-Μπομπίνσκα «Ο ρόλος πολιτικής συνοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής» και έκθεση Εστάρας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, Υλοποίηση και Εφαρμογή. Δίνω το λόγο στον εισηγητή κύριο Κοτσολίνο για τέσσερα λεπτά. Η έκθεσή μου θέτει ως στόχο να θέσει στο στόχο της μελλοντική πολιτικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής το ζήτημα των πόλεων και του αστικού ευρωπαϊκού ιστού. Γιατί μπορούν να αποτελέσουν οι πόλεις μια πάρα πολύ σημαντική ε, πλατφόρμα προκειμένου να δοθεί μια οικονομική ανάκαμψη καθώς επίσης και προώθηση των θέσεων εργασίας. Το ζήτημα των πόλεων και των αστικών περιοχών αποτελεί μια πολύ σημαντική πρόκληση για το μέλλον. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει στις πόλεις μία μείωση του πληθυσμού, γύρανση του πληθυσμού. Έχουμε φαινόμενα μιας νέας ένδυας, κοινωνικής και οικονομικής ένδυας. Η πόλη όμως από την, από την άλλη και ο αστικός ιστός μπορούν να αποτελέσουν κέντρο δημιουργικότητας, ευφυΐας, μπορούν να δημιουργήσουν πολλές διαφορετικές εμπειρίες στη συνύπαρξη πολλών διαφορετικών εθνικοτήτων. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για τις πόλεις. Ένα σχέδιο για τις αστικές περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα χρησιμοποιούνται τα νέα μέσα που προβλέπονται από τα Ελευθερωτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. Ένα σχέδιο το οποίο θέτει συγκεκριμένους στόχους, στους οποίους προσπαθούν να τονίσω στα πλαίσια της έκθεσής μου. Ένας στόχος είναι η αναβάθμιση των προαστίων. Ένα πραγματικό πρόγραμμα για να έχουμε μια καλύτερη κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση των πόλεων. Επίσης, μια καλύτερη οικονομική αποδοτικότητα των βιομηχανικών κτηρίων καθώς επίσης και των κατοικιών. Ως προς αυτό θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα επίσης, ένα σχέδιο για την ασφάλεια, τη διασφάλιση της αστικής μας και στεγαστικής κληρονομιάς. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα φαινόμενα, όπως οι κλιματικές αλλαγές, ή το ζήτημα της ειρηνικής συνύπαρξης στις αστικές περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την προστασία ορισμένων πόλεων οι οποίες πλήττονται από σεισμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε ολόκληρες περιφέρειες της Υπήρου μας. Χρειαζόμαστε επίσης ένα σχέδιο για κάποιες νέες κοινωνικές κατοικίες είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι πάρα πολλά κράτη-μέλη έχουν εγκαταλείψει οποιαδήποτε πολιτική που θα μπορούσε να υποστηρίξει τι κοινωνικέ κατοικίε. Μάλιστα, αυτό που βλέπουμε σε πάρα πολλέ χώρε είναι ότι γίνεται ακριβώ το αντίθετο. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξαρτώμαστε μόνο από τις δυνάμεις της αγοράς προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες αστικές υποδομές, ιδίως αυτές οι οποίες θα πρέπει να προστατεύσουν τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι νέοι και οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι. Επίση, υφίσταται ένα πάρα πολύ άλλο σημαντικό ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με τι πόλει και τον αστικό δίκτυο. Αυτό έχει να κάνει με την κινητικότητα των ανθρώπων, των προϊόντων και των υπηρεσιών. Θα μπορούσαμε ω προ αυτό να πούμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα και για το ζήτημα της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος. Τέλος υπάρχει και το ζήτημα της ε, διατήρησης της ιστορικής κληρονομιάς των πόλεων μας. Εδώ πραγματικά έχουμε έναν τεράστιο πλούτο που καλούμεθα να προστατεύσουμε και μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη την οικονομική. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και κάποια παλιά προβλήματα τα οποία εντάσσονται σε αυτή τη νέα πρόκληση. Να καταφέρουμε να δούμε τι θα γίνει με τι περιοχέ που βρίσκονται στι παρυφέ των πόλεων, με τα προάστια. Ένα τεράστιο, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ουσιαστικά χρειαζόμαστε μια αστική πολιτική η οποία θα μειώσει την χρήση τη υπαίθρου ή την επέκταση των πόλεων στην Ήπεθρο. Το ζήτημα αυτό ε, έχει λάβει πάρα πολύ δραματικά φαινόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεσή μου αναφέρομαι και σε δύο ακόμα παρατηρήσεις. Ένα 5% των κονδυλίων που θέλουμε να δώσουμε στις ε, πολιτικές ε, ανάπτυξης των πόλεων θα πρέπει να ενταχθούν στο νέο προγραμματικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε μια πιο ισχυρή νομική βάση όσον αφορά το ζήτημα της αντιμετώπισης των πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε καλύτερες πολιτικές. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο επόμενος εισηγητής, ο κύριος Βάογκαν, για τέσσερα λεπτά. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπω ότι ο Επιτρόπος είναι εδώ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δόθηκε να κάνω αυτή την έκθεση, γιατί νομίζω ότι η πολιτική συνοχή είναι ζωτική ε, για τι περιοχέ Ευρώπη, αλλά και ελπίζουμε να έχουμε στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Δεν είναι όμω η χρηματοδότηση το μόνο ε, στοιχείο. Θα πρέπει να υπάρχουν και οι σωστοί κανόνε, κανονισμοί για την πολιτική συνοχή για να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και απασχόληση. Χαιρετίζω λοιπόν ιδιαίτερα τι προτάσει τη Κομισιόν για, τον, για τους κανονισμούς και ιδίως ε, τις προτάσεις ε, για ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για πέντε από τα μεγαλύτερα ταμεία. Αυτό θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, να βελτιώσουμε την απλούστευση για τους ετούντες ε, και να έχουμε και καλύτερη, ευκολότερη πρόσβαση των ετούτων σε διάφορα ευρωπαϊκά κονδύλια και ταμεία. Όταν οι κανονισμοί πρωτοπροτάθηκαν, φάνηκε να υπάρχει ελλειπές επίπεδο λεπτομέρειε για τη δημιουργία μηχανισμών για τη συνένωση των πέντε ταμείων. Έχουμε τώρα κάποιε προτάσει για συμφωνητερική σχέση, προτάσει για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, προτάσει ε, για κώδικα διοντολογία, ε, για κοινά σχέδια δράση, ε, για πρωτοβουλία τοπικών ε, κοινοτήτων, εδαφική, ολοκληρωμένε εδαφικέ επενδύσει. Όλα αυτά είναι καλέ ιδέε και θα πρέπει να τι καλωσορίσουμε, να τι επικροτήσουμε όλε. Αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται, κατά την άποψή μου, είναι οι μηχανισμοί ώστε όλα αυτά ε, να. Ε, οδηγήσουν στη συνένωση των ταμείων που εξέγησα προηγουμένως. Ήρθα λοιπόν σε διαβουλεύσεις με πολλούς ε, ενδιαφερομένους ε, φορείς από όλο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα συζητήσει στρογγυλής τραπέζης, ε, με επαγγελματίες, με πλεκομένους φορείς τοπικές αρχές που έχουν καθημερινή επαφή και ενασχόληση με αυτά τα προγράμματα και πιστεύω ότι ξέρουν τι πρέπει να κάνουμε για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, για το μέλλον. Και Ιδίω αυτή η στρογγυλή τράπεζα ήταν πάρα πολύ σημαντική και χρήσιμη γιατί καταφέραμε να διερευνήσουμε κάποιου μηχανισμού για τη συνένωση αυτών των ταμείων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ένα καλό παράδειγμα ήταν η Ουαλία. Και βέβαια ε, φαντάζομαι ότι θα το περιμένατε από μένα σας ένα τέτοιο παράδειγμα. Γιατί στην Ουαλία ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μετά το 2014 μία ενιαία δικτυακή πύλη. Να έχουμε ενιαία δηλαδή αίτηση, πληρωμή και διαδικασία παρακολούθησης. Μοναπευθετική θηρίδα αν θέλετε σχεδόν για τους ετούντε και για την διαχειριστική αρχή. Ένα άλλο καλό παράδειγμα ήταν στις κατοχώρες όπου κονδύλια διαφόρων προγραμμάτων θα ε, δοθούν ε, στις τοπικές αρχές για να μπορέσουν να δημιουργήσουν δέσμες, ε, πακέτα κονδυλίων για να χρηματοδοτήσουν τοπικά ε, project. Στο Μάντσεστερ επίσης έχουμε ένα πρόγραμμα όπου υπάρχει ένα, μια πρόταση για ένα ETI που θα έχει τη χρηματοδότηση ε, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από άλλες πηγές. Παραδείγματο χάρη θα προτείνουν ένα σχέδιο υποδομής ε, χρησιμοποιώντας ταμεία του ΕΤΠΑ και χρησιμοποιώντας ταμεία του ΕΚΤ για την εκπαίδευση αυτών που θα ασχοληθούν με αυτό το project και αυτό το επεξεργαζόμαστε ως μια πρόταση για μετά το 2014. Και βέβαια θα υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα από ε, περιφέρειες ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε κατά την άποψή μου είναι να συλλέξουμε όλε αυτές τις ιδέες και τις καλε πρακτικές και να βρούμε τρόπου ε, ανταλλαγή των καλών πρακτικών αυτών σε ολόκληρη την επικράτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίτροπε, εύχομαι να ακολουθήσετε τι συστάσει και τι προτάσει μα ε, από αυτή την έκθεση τη πρωτοβουλία, ώστε τελικά να βρούμε τρόπου, μηχανισμού, ώστε τι ιδέε αυτέ, τι καλέ αυτέ ιδέε να τι κάνουμε πράξη. Η τοπική ε, κοινωνία, οι τοπικέ αρχέ να μπορέσουν να συνενώσουν κονδύλια των μεγάλων ταμείων για να χρηματοδοτήσουν μεγάλα project. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο και για να διασφαλίσουμε μεταξύ άλλων ότι θα επιτύχουμε τους στόχους για την Ευρώπη του 2020 και είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος ε, να έχουμε μεγαλύτερη οικονομική ευημερία στις περιοχές ε, και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η επόμενη εισηγήτρια Κολάρσκα Μπομπίνσκα για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία να πετύχουμε συνέργειες μεταξύ περιφερειακής πολιτικής και ενεργειακής πολιτικής. Είναι μια ευκαιρία ταυτόχρονα διτά για να ανταποκριθούμε στους στόχους αμφωτέρων αυτών των πολιτικών και να βελτιστοποιήσουμε τις δράσεις μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαντικά κονδύλια έχει επιμερίσει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης όσον αφορά και τα ενεργειακά θέματα για την ενεργειακή πολιτική. Τώρα πρέπει αυτά τα κονδύλια, αυτούς τους πόρους να, το, να τους χρησιμοποιήσουμε με, με τους βέλτιστους τρόπους. Γι' αυτό καθίσταστε σαφές ότι σε σχέση με τα κονδύλια που θα χρηματοδοτήσουν τι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής, πρώτιστα θα πρέπει να παράσχουν υποστήριξη για την περιφερειακή ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να βοηθήσουν έτσι να αμβληνθούν, να καλυφθούν οι παρεκκλήσεις και οι διαφορές και οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης. Το να βελτιώσουμε τα θέματα ενεργειακού ανεφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει κίνητρα και να δώσει ερεθίσματα να καλύψουν τη διαφορά που τις ε, χωρίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις επενδύσεις σε αποκεντρωμένες δράσεις μέσω ειδικών κονδυλίων. Καθίσταται σαφές από την έκθεση ότι κύριοι στόχοι της περιφερειακής πολιτικής και της ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει να εμπεριέχουν τις επενδύσεις που είναι αναγκαίες στους ενεργειακούς πόρους αλλά και την ενεργειακή αποδοτικότητα στις επιδόσεις μας στην εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας όσον αφορά και τις επενδύσει στις υποδομές. Πολλέ φορέ κάνουμε λόγους, λόγο για πηγές ενέργειας, όμω ε, δεν αναφερόμαστε τόσο συχνά στα θέματα διαβίβαση, μεταφοράς ενέργειας από την πηγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Πολλά μπορούν να γίνουν για το δίκτυο διαβίβαση μεταφοράς ενέργεια και όσον αφορά και τι υποδομές γενικότερα. Πολλά μπορούν να βελτιωθούν. Τούτων λεχθέντων, οι περιφέρειες της Ευρώπης είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Δεν μπορούμε ισοπεδωτικά να δράσουμε με μία δράση που θα αφορά όλες τις περιφέρειες. Δεν θα είναι θετικό αυτό. Υπάρχουν περιφέρειες και περιοχές που επιθυμούν να, να ενισχύσουν με τις επενδύσεις ε, στον εξυγχρονισμό των κτηρίων. Ε, άλλες ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μεταφορά, στο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας όλοι αυτοί οι στόχοι, αυτό το οποίο έχουν κοινό ως στοιχείο, ως κοινό παρονομαστή είναι ότι είναι ευρωπαϊκοί στόχοι. Και μια και έχουν διαφορές οι περιφέρειες και οι περιοχές όσον αφορά το επίπεδο ανάπτυξής τους, καθιστά σαφές η έκθεση ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να έχουν λόγο που μπορούν να αρθρώσουν όσον αφορά τα αιτήματά τους σε σχέση με τα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι περιφέρειες, οι περιοχές τι πρέπει να επιδοτηθεί και να, πού θα υπάρξουν επενδύσεις, ποια κονδύλια, ποια ποσά θα επενδυθούν, πού και για ποια χρήση και σκοπό. Δεν θέλουμε να υπάρξει διασπάθηση ή απώλεια κονδυλίων. Δεν είναι μόνο το θέμα της δαπάνης κονδυλίων, είναι της βέλτισης δαπάνης ε, και χρήσης κονδυλίων για περιοχές και περιφέρειες για παράδειγμα που συγχρονίζουν ε, τα σχολεία τους ή για τέτοιες δράσεις θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι η περιφέρεια, η περιοχή που έχει κάνει τα του οίκου τη και έχει κάνει σωστά τη δουλειά της δεν θα πρέπει να υποστεί κυρώσεις και στην επόμενη ε, στις επόμενες ε, προοπτικές, δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για τα θέματα ενέργειας. Όμως ε, η περιφερειακή πολιτική δεν μπορεί να υφίσταται τις θυσίες και τις περικοπές όταν έρχεται η ώρα και η στιγμή υλοποίησης ενός προγράμματος. Η πολιτική συνοχή δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο για την σωστή χρήση και την αποτελεσματική χρήση κονδυλίων. Καλό θα ήταν να το θυμόμαστε και να το επαναλαμβάνουμε αυτό ως αρχή. Η πολιτική συνοχή πρέπει να υφίσταται, να λειτουργεί, να επιτυγχάνει, να υλοποιεί του στόχου τη. Μπορεί να διασυνδέεται με άλλε πολιτικέ, όμω πρέπει να έχουμε ξεχωριστέ πηγέ χρηματοδότηση για την επίτευξη του κάθε στόχου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σταράσα έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το 2002 δημιουργήθηκε το Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανταποκριθεί σε φυσικές, σοβαρές φυσικές καταστροφές που έπληξαν κράτη-μέλη ή ε, χώρες ε, που ήταν στη διαδικασία προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει κανένα άλλο εργαλείο ε, μέχρι στιγμή ε, πλην αυτού που παρεμβαίνει σε περίπτωση καταστροφών. Αυτά τα 10 χρόνια ήταν ε, επιτυχημένα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Ταμείου. Η αρχή τη Αλληλεγγύη Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη χάρη στο Ταμείο αυτό μια αρχή η οποία πήρε σαρκα και ωστά. Όμω αυτά τα 10 χρόνια επίση μπορέσαμε με την εμπειρία μας να δούμε ακριβώς τι αδυναμίες είχε αυτό το ταμείο, τι ελλείψει. Είδαμε ότι οι σοβαρές φυσικές καταστροφές ε, που δημιουργούν ε, ένα, ε, μια βλάβη μεγαλύτερη από το κατόφλι για την παρέμβαση λειτουργήσαν σχετικά καλά. Όμως είδαμε ότι σε ό,τι αφορά περιφερειακές καταστροφές που αλλάζουν δηλαδή τις συνθήκες σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια και επηρεάζουν την καθημερινότητα ε, των ανθρώπων, ε, τις συνθήκες διαβίωσής τους και επηρεάζουν ε, για μακρόχρονικό διάστημα την κατάσταση. Είδαμε τις προκειμένες αυτές περιπτώσεις πολλές αιτήσει κατατέθηκαν από τις περιφέρειες, όμω δεν έγιναν δεκτέ. Πάνω από το 60% των αιτήσεων για τέτοιες καταστροφές ε, έγιναν και επειδή ήταν ασαφής η έννοια, ε, δεν ήταν σαφείς οι δείκτες, πολλές προσδοκίες μεν δημιουργήθηκαν ε, από την πλευρά των περιφέρειων, αλλά τελικά δεν έγιναν δεκτές οι αιτήσει τους. Σήμερα λοιπόν ε, στόχος μας και με την έκθεση που υποβάλλουμε είναι να διορθώσουμε την κατάσταση αυτή, την αοριστία δηλαδή ε, σε σχέση με αυτές τις φυσικές καταστροφές, τις περιφερειακές. Αυτά τα 10 χρόνια κάτι άλλο που είδαμε είναι ότι θα μπορούσε να γίνει πιο ευέλικτο και πιο γρήγορο το ταμείο αυτό. Δηλαδή από τη στιγμή που έχουμε μια καταστροφή μέχρι τη στιγμή που εισπράττει ε, τα χρήματα το κράτος μέλος μπορεί να περάσουν 9 με 12 μήνες και αυτό σίγουρα είναι πολύ σοβαρό για τους πληγέντες περιοχής. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια απλούστευση των διαδικασιών του Ταμείου να είναι πιο γρήγορες, ε, πιο απλές και να δίδονται και κάποιε προκαταβολικές πληρωμές. Είδαμε επίση ότι σε αυτές τις λεγόμενες βραδίες καταστροφές, παραδείγματος χάρη ξηρασία, ε, το, η προθεσμία 10 εβδομάδων ε, για να υπάρξει εκτίμηση των ζημιών δεν είναι δυνατό να τηρηθεί. Σε τέτοιες βραδίες λοιπόν καταστροφές θα μπορούσε να είναι πιο ευέλικτο το Ταμείο. Τέλος, πρέπει να πω ότι ζητήσαμε μια μεταρρύθμιση του κανονισμού, αλλά χωρίς σε καμία περίπτωση να θίξουμε τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, ε, τις δαπάνες ή τα κριτήρια της επιλεξιμότητας για επιδότηση. Θα θυμάστε ότι πρόσφατα, κάποια χρόνια πριν, είχε γίνει μια πρόταση που δεν έγινε δεκτή από το Συμβούλιο γιατί αφορούσε τι ε, δαπάνε, το κόστο και δεν τη δέχθηκε το Συμβούλιο. Και μάλιστα έλεγε ότι πέραν των φυσικών καταστροφών έπρεπε να συμπληρωθούν και άλλε καταστροφέ. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ε, το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε να προχωρήσει η έκθεση. Το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θέλουμε να δώσουν το πράσινο φω, άρα δεν θίγουμε σε καμία περίπτωση ούτε τα, πάνη, ούτε τα κριτήρια ε, επιλεξιμότητα για να δοθεί μια επιδότηση. Στην περίπτωση των περιφερειών, επαναλαμβάνω, προτείνονται κριτήρια όπω το καθάριστο εγχώριο προϊόν για να έχουμε ένα παρκέ κατόφλι που θα είναι προσαρμοσμένο στην περιφέρεια που θα κάνει την αίτηση. Επίση, ζητάμε να απλουστευθούν όλες οι διαδικασίε και σε κάποιες περιπτώσεις, με παραδείγματι η Κομισιόν μέχρι τώρα, Είχε μια πράξη παραχώρησης και μετά ε, γινόταν πιο συγκεκριμένοι οι όροι ε, για την επιδότηση. Θέλουμε να, όλα να γίνουν μία, σε μία νέα πράξη. Θέλουμε λοιπόν να είναι πιο αποτελεσματικό, πιο διαφανές το τομέα και νομίζουμε ότι με την προτάσει μα θα το πετύχουμε. Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος, ο Επίτροπος Χάννα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, καταρχήν θα ήθελα και εξ ονόματος ε, του συνόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ευχαριστήσω τις εισηγήτρες και εισηγητές για τις ε, ε, πολύ καλές εκθέσεις τους. Δεδομένου του ότι βρίσκονται υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, αυτές οι εκθέσεις συνεισφέρουν με ένα σημαντικό τρόπο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της εδαφικής συνοχής των αστικών κέντρων και περιοχών και να μπορέσουμε να διοργανώσουμε την ενεργειακή μας πολιτική με τον καλύτερο τρόπο. Η ευρεία υποστήριξη που έτυχαν αυτές οι εκθέσεις στις κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι ένα σημαντικό μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και χαίρομαι για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ευθυγραμμίζονται προς κοινή κατεύθυνση. Η περιφερειακή αυτή διάσταση, η συνιστόσα για την πολιτική μας έχει τεράστια σημασία. Ο κύριος ε, Κοσολίνο υπογραμμίζει την, ε, ο κύριος Κοσολίνο υπογραμμίζει την διασύνδεση μεταξύ αστικών κέντρων και των περιφερειών για την υλοποίηση της ε, αναβάθμισης των στόχων μας και για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης 2020. Είτε πρόκειται για την ενίσχυση της καινοτομίας, οι πόλεις διαδραματίζουν ένα ξεχωριστό ιδιαίτερο ρόλο και πρέπει να εντάσσονται σε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό είναι απαραίτητο απαραίτητο για μένα υπό την πολυσχηδή διακυβέρνηση και διαχείριση και το επαναλαμβάνω αυτό θα τονίσουμε το θέμα στις διαπραγματεύσεις ώστε οι κυβερνήσεις να λαμβάνουν υπόψη και το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αυτών των συνιστοσών στην εκπόνηση των πολιτικών τους. Όπως είπαμε, σχεδιασμός και υλοποίηση στο δυνατόν ευρύτερο πλαίσιο πρέπει οι εμπλεκόμενοι να είναι εταίροι και οι πόλεις, αλλά πρέπει να εκπονήσουν και να δημιουργήσουν τα αναγκαία μέσα και εργαλεία. Παραμένουμε σε αυτό το αίτημα. Τουλάχιστον 5% των κονδυλίων θα πρέπει για τέτοια ολοκληρωμένα προγράμματα αστικών κέντρων να χρησιμοποιούνται που θα διαμορφώνονται από τα ίδια τα αστικά κέντρα, από τις ίδιες τις πόλεις. Και έτσι αυτό το 5% να αναφέρεται στην ολοκληρωμένε στις ολοκληρωμένες περιφερειακές πρωτοβουλίες. Φυσικά πέρα από αυτό, κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη θα διατίθενται και στο μέλλον για την, όπως και σήμερα συμβαίνει, για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Τονίζεται στις εκθέσεις αυτές ότι με μια κοινή στρατηγική δημιουργείται, πρέπει να δημιουργηθεί ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Η εταιρική σχέση θα διαδραματίζει ως εργαλείο ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την διαμόρφωση και υλοποίηση των πολιτικών αυτών σε αυτές τις περιοχές στο επίπεδο των κοινοτικών, ε, της κοινοτικής εκπροσώπησης ε, των τοπικών αρχών ε, και του επίπεδου των Δήμων και ε, Κοινοτήτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο με οδηγίε για τη δράση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής μπορώ να σα διασφαλίσω ότι με μέγιστο ζήλο εργάζεται η Γενική Διεύθυνση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δυνατόν γοργότερα θα, θα υπάρξουν κατευθυντήρε γραμμέ που θα δοθούν ε, για να υποστηριχθούν οι εμπλεκόμενοι. Θα πρέπει να στρέψουμε περισσότερο το βλέμμα και στο διοικητικό δυναμικό. Έχουμε κοινή ευθύνη με τα κρατη να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια αυτά θα χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποβαίνουν προ όφελο τη απασχόληση και τη ανάπτυξη. Αυτό ισχύει φυσικά και για την αηφόρο ενεργειακή πολιτική που η κυρία Κοράσκα Μπομπίνσκα πιο πριν με την έκθεσή τη ανέφερε και μπορώ να διασφαλίσω ότι μέσω των μέτρων για την πολιτική συνοχή σε συνδυασμό με την ενεργειακή πολιτική συμμερίζομαι τι τοποθετήσει και του προσανατολισμού τη. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένε δράσει ώστε προς αυτή την κατεύθυνση στις επιμέρους περιφέρειες και περιοχές να δραστηριοποιηθούμε όπως πρέπει, όπως για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ολοκληρώνοντας θέλω να πω κάτι για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Στα 10 χρόνια της ύπαρξης από το 2002 ε, στο 2012 και σε σχέση με την δημιουργία διάθεσης κονδυλίων 3,1 δις ευρώ μπορέσαμε να βοηθήσουμε. Η Ευρώπη είναι μια κοινότητα αλληλεγγύη. Ε, που μπορούμε να πούμε ότι με το Ταμείο Αλληλεγγύης ε, έχουμε και ένα αντίστοιχο μέσο για να δράσουμε αποτελεσματικά. Είμαι πεισμένος ότι αυτό το μέσο ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο αποτελεσματικά μπορούμε να το πρικοδοτήσουμε και να το ενεργοποιήσουμε ευχαριστώ για την ε, αντιμετώπιση σε σχέση με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε σχέση με το Ταμείο Αλληλεγγύης. Στο άμεσο, στο εγγύς μέλλον θα υποβάλουμε μια νομική πρόταση σχετικά και ήδη σήμερα ζητούμε την υποστήριξή σας σε, αυτό το, σε αυτή την πρωτοβουλία μας. Ευχαριστώ και πάλι για την εξαιρετική εργασία και συνεργασία που είχαμε ώστε να μπορέσουν αυτά να ευδοκιμήσουν και κυρίως θα πρέπει οι Δήμοι κοινότητα στο περιφερειακό επίπεδο να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν. Χρειαζόμαστε το βέλτιστο πλαίσιο υποστήριξη. Πρέπει να υπάρξει συνάφεια, συνεκτικότητα και συνοχή σε σχέση με αυτέ τι δράσει με τα μέσα και εργαλεία που έχουμε δημιουργήσει, ώστε οι εμπλεκόμενοι στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ακόμα καλύτερα να μπορούν να καλυφθούν στι ανάγκε του και τα αιτήματά του, Και έτσι όπω και στο παρελθόν, έτσι και στο μέλλον θέλω να ε, είσαστε ισχυρό εταίρο εσεί ω Ευρωβουλή έναντι ημών της Ευρωπαϊκής Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Ισμενόβα, εξ ονόματος Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, η εδαφική συνοχή αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση του κυρίου Βόγκαν αποτελεί μια πολύ καλή βάση προκειμένου να εκπονηθεί μια στρατηγική και να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Θα χρησιμοποιηθεί λοιπόν το κοινό αυτό στρατηγικό πλαίσιο προκειμένου να εφαρμοστούν καλύτερα επιτόπου τα ταμεία, τα κονδύλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τελικά τις τοπικές κοινότητες. Η προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω θα πρέπει ενεργώς να εφαρμοστεί με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στην, στο προγραμματισμό της στρατηγικής για την τοπική ανάπτυξη. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητα και θα πρέπει να μειωθεί το διοικητικό άχθος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εξ ονόματος Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας, ο κύριος Έντσου έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να κατανοήσουμε το εξή. Η πολιτική συνοχή έχει θεμελιώδη αξία και σημασία για το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι από την επιτυχία τη θα εξαρτηθεί η προαγωγή των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών και μάλιστα προ όφελο όλων των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην περικοπούν, να μην διαγραφούν τα κονδύλια για την πολιτική συνοχή κατά το επόμενο διάστημα. Έχω συντάξει μια γνωμοδότηση από πλευρά τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Λέγω, τα, τα ταμεία αυτά από πλευρά τη διαθροτική πολιτική πρέπει να συνεχίσουν να έχουν θετικά αποτελέσματα στι λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχέ, κυρίω στην Ανατολική Ευρώπη, όπου υπάρχουν πολλέ ελλείψει και μειονεξίε για την εξυγίαση κτηρίων και αλλού. Πρέπει να υποστηρίξουμε τέτοιε δράσει μέσω μέσων, χρημα... Ε, μέσω, μέσων ε, δράση και πρωτοβουλία και μέσων εγγύηση. Χρειαζόμαστε ιδιαίτερε προτεραιότητε για τι υποδομέ. Σε σε, ιδιαίτερο βαθμό και τρόπο. Εδώ η ολοκλήρωση, η διασύνδεση των κονδυλίων των διαθετικών ταμείων με τη διευκόλυνση της διασύνδεσης για την Ευρώπη πρέπει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Ξεκινώντας ε, τώρα από τις ε, κοινοβουλευτικές ομάδες, ο κύριος Ματσόνη. Δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρία Ματσόνη, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για το έργο που επετέλεσαν και το αντικείμενο των εκθέσεων αυτών εξειδικευμένα στο πλαίσιο αυτής της κοινή συζήτησης ε, που διεξάγεται στην Ολομέλεια. Τον στόχο που έχουμε ενώπιόν μας ε, να υπάρξει μεγαλύτερη κοινωνική συνιστόσα στην πολιτική συνοχή ε, πρέπει να τονίσουμε ότι η σημασία είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε αυτές τις τέσσερις εκθέσεις και αναγνωρίζεται από τον Επίτροπο Χάν ότι υπάρχει κοινή προσπάθεια και κοινή ευθυγράμμιση προς κοινέ κατευθύνσει και προσανατολισμούς. Ο κύριος Κοτσολίνο θα ήθελε οι πόλεις να βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής συνοχής. Όχι όμως οι πόλεις χωρίς περίγυρο και χωρίς ε, τις ε, συνοικίες και την ε, ε, γύρω τους περιοχή, αλλά με αυτή την περιοχή και τις ε, γύρω τους. Μπορούν να γίνουν ένας κινητήριος μοχλός και αυτό θα πρέπει να γίνει με οικοσυμβατό τρόπο στα πλαίσια της ανάπτυξης των πόλεων χρησιμοποιώντας κάποια μέσα όπως το μέσο της αλληλεγγύης με στοχευμένο και πιο αποτελεσματικό από ό,τι μέχρι τώρα τρόπο. Αυτό το μέσο θα πρέπει να έχει κάποιες δυνατότητες χρήσης πιο εύκολες, πιο χρηστικές από αυτό το οποίο μας έδειξε η εμπειρία των προηγούμενων ετών. Σαν σκιώδης εισηγήτρια της εκθέσεως Κοτσολίνο, εγώ έχω συγκεντρώσει την προσοχή μου σε θέματα όπως οι στόχοι της συγκεκριμένης έκθεσης. Και είδα ότι σε συνεργασία στενή με τον εισηγητή προσπαθήσαμε να δώσουμε και στη διάσταση των περιοχών των πόλεων ε, μια υπογράμμιση που απαιτείται από την συγκυρία. Οι στόχη της ανάπτυξης των πόλεων συνδέονται, αγκυρώνονται με τις προοπτικές που έχουμε για το 2020. Και το 5% των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το ελάχιστο δυνατό, όχι το μέγιστο για την ανάπτυξη των πόλεων, των αστικών περιοχών. Θα πρέπει στα πλαίσια του προγραμματισμού να εμπλακούν οι τοπικοί άρχοντες, στα πλαίσια ενός συμμετοχικού σχεδίου και στη φάση της λήψης απόφασης και όχι μόνο στη φάση της κατανομής των πόρων. Ευχαριστώ πολύ. Χριστιανοδημοκράτες Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πολιτική συνοχή είναι πραγματικά ένα πολύ ευρύ πεδίο. Και αυτό φαίνεται και από τη συζήτηση εδώ, από την αστική ανάπτυξη, τη συμβολή των πόλεων την οικονομία, ε, μέσω της εδαφικής ανάπτυξης και της εδαφικής συνεργασίας μέχρι την ενεργειακή πολιτική και την συμβολή της ε, ενεργειακής πολιτικής στην πολιτική συνοχή μέχρι το Ταμείο Ελεγγύης. Και θα μπορούσα να σας αναφέρω και άλλα θέματα που συμπεριλαμβάνονται εδώ. Κατ' ουσία πρόκειται για, ένα, για μια πολύ θετική εικόνα, αλλά θα πρέπει εδώ να είμαστε και λίγο προσεκτικοί, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό εδώ να θέσουμε ξεκάθαρους στόχους για την πολιτική συνοχή και να αξιοποιήσουμε τα διαθέσιμα οικονομικά κονδύλια επικεντρώνοντάς τα σε αυτούς τους στόχους. Ε, δεν γίνεται να ξοδεύουμε χρήματα βάσει αρχής των συγκοινωνών δοχείων, όπως το κάναμε στο παρελθόν. Αυτό το προσανατολισμό της ε, πολιτικής ε, συνοχής μπορούμε να τον ε, παρακολουθήσουμε, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ένα ευρύτερο πεδίο, δηλαδή τη δική μας ε, ε, εργασία προβολής προς την κοινή γνώμη σε σχέση με την πολιτική συνοχή γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί να αυξηθεί η αποδοχή, ο βαθμός αποδοχής της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και αυτό μπορεί να το πετύχουμε εάν λάβουμε σοβαρά την αρχή της εταιρικής συνεργασίας και λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τους τοπικούς εταίρους. Μόνο στην περίπτωση αυτή θα στεφθούν με επιτυχία τα προγράμματα. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα την ευρωπαϊκή πολιτική εντός της πολιτικής συνοχής, αλλά και σε σχέση με άλλες πολιτικές. Και τέλος θα πρέπει να πούμε ότι ε, δεν θα χρησιμεύσει τίποτα μια καλά σχεδιασμένη πολιτική εάν δεν επαρκούν τα κονδύλια. Θα πρέπει να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στη διαπραγματεύση με το MSF, ούτως ώστε να μπορέσουμε να χαράξουμε μια θετική πολιτική για τους πολίτες της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τους φιλελεύθερους. Η κυρία Μανέσκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτή την έκθεση. Τα μέτρα και οι δράσει οι οποίε ε, προτείνονται εδώ βεβαίω έχουν σαν στόχο την πολιτική συνεχίση και το ζητούμενο εδώ είναι μέσα των διαφορετικών ταμείων να μπορέσουμε να το πετύχουμε ε, το ταχύτερο δυνατό να ανακάμψει η οικονομία. Ιδιαίτερα σημαντικέ εδώ είναι οι πόλει, γιατί στα, τα κέντρα αστικοποίηση πλήττονται σοβαρά από την κρίση και εδώ ανακύπτουν πολύ σοβαρά προβλήματα, ανεργία, διακρίσεις, φτώχεια. Και θα πρέπει να σκεφτούμε το ρόλο κλειδί που παίζουν εδώ οι πόλεις. Και εδώ οι στόχοι της Ατζέντα 2020 είναι σημαντικοί, καθώς και οι στόχοι. Ε, θα μπορέσουμε να αφήσουμε την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα παγκοσμίω μόνο εφόσον αξιοποιήσουμε το δυναμικό της αστικής ανάπτυξης αλλά συνδέσουμε και στην ανάπτυξη των περιφερειακών κέντρων. Και εδώ είναι σημαντικό να προωθήσουμε επενδύσει στον τομέα τη ενέργεια, των υποδομών και σε δράσει που βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και αυτό είναι σημαντικό για την περιφερειακή ανάπτυξη. Τα διαθετικά ταμεία έχουν να παίξουν ένα ρόλο κλειδί, ιδιαίτερω για την επίτευξη αυτών των στόχων και είναι πολύ σημαντικό για την επόμενη προγραμματική περίοδο και θα πρέπει να μερμνήσουμε ότι όσο στο επίπεδο τη Επιτροπή να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, ούτω ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά απορρόφηση αλλά να δοθούν και τα αναγκαία κονδύλια. Ε, χρειαζόμαστε απλές διαδικασίες, ξεκάθαρες διαδικασίες προκειμένου να μειωθεί ο βαθμός γραφειοκρατίας και να εξηγιανθούν οι διοικητικοί μηχανισμοί. Επίσης είναι σημαντικό να συμμετάσχουν οι περιφερειακές και τοπικέ αρχές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και να εξασφαλιστεί και ένας μεγάλος βαθμός ευελιξίας. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των Πρασίνων, ο κύριος Χρυσόγελος για ένα λεπτό. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελεγγύης ξεκίνησε αμέσως μετά τις πλημμύρες του 2002. Ε, η κλιματική αλλαγή όμως και άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις έχουν οδηγήσει σε αύξηση της συχνότητας και της έντασης των ε, φυσικών καταστροφών. Το 2005 το Συμβούλιο μπλόκαρε τις αλλαγές στο Ταμείο. Αυτή τη φορά πρέπει να γίνει δεκτή από το Συμβούλιο η πρόταση επιτροπή με τις τροπολογίες του Ευρωκοινοβουλίου, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του Ταμείου με δεδομένη την αύξηση συχνότητας και της έντασης των φυσικών καταστροφών και στην Ευρώπη. Από το 1980 στο 2011 οι συνολικές ζημιές στον ευρωπαϊκό χώρο από υδρολογικά, γεωφυσικά, κλιματολογικά και ακραία φαινόμενα έφτασαν τα 455 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι φυσικές καταστροφές προκάλεσαν 110.000 θανάτους. Οι ασφάλειες κάλυψαν μόνο το 27% των περιπτώσεων, ενώ δεν καλύπτουν συνήθως πολλά από τα φαινόμενα τα καταστροφικά το ταμείο λοιπόν πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο στην αποτελεσματική αποκατάσταση περιοχών και της κοινωνικής ζωής σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αλλά η συνεισφορά του ταμείου πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα βελτιώνει τις πολιτικές και πρακτικές πρόληψη των φυσικών καταστροφών καθώς και θα περιορίζει τι συνέπειε του ο καλύτερο τρόπο φυσικά και πιο οικονομικό για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών είναι η πρόληψη. πρέπει όμω να βελτιωθεί και η διαδικασία να είναι πιο ξεκάθαρε οι περιπτώσει που μπορούν να στηριχθούν από το ταμείο μια και το 60 των αιτήσεων απορρίφθηκε στην προηγούμενη περίοδο να απλοποιηθούν οι διοικητικέ γραφειοκρατικέ διαδικασίε να βελτιωθεί ο χρόνο που απαιτείται μέχρι να φτάσουν οι οικονομικοί πόροι από του ευρωπαϊκού θεσμού στα κράτη μέλη αλλά και τα κράτη μέλη στου δικαιούχου των αποζημιώσεων στι Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των Ισιάρο, ο κύριος Φλάσακ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, γνωρίζουν όλοι ότι τα θέματα τα οποία συζητούμε ε, τώρα είναι σαφώς και ε, άρρηκτα συνδεδεμένα με την πολιτική συνοχή, καθώς επίσης ε, και με το δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2020 θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι σαν να μην, σαν να μην συζητούσαμε τίποτα γιατί διαφορετικά ε, δεν θα μπορέσουμε να γυρίσουμε στις πατρίδες μας ε, και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους, ε, τις συνθήκες αυτές βάσει των οποίων θα χρησιμοποιηθούν σωστά και μέχρι το 2020 όλοι οι πόροι των ταμείων. Οι πόλεις βεβαίως θα πρέπει να παίξουν πολύ πιο σπουδαίο ρόλο στο μέλλον. γιατί είναι λίγες ακόμα οι πόλεις αυτές οι οποίες έχουν την δυνατότητα ε, να διαχειριστούν καλά τους πόρους τους. Όμως μόνο οι πόλεις οι οποίες είναι σε θέση να διαχειρίζονται σωστά τις, τους πόρους τους θα μπορέσουν ε, να προχωρήσουν και να προοδεύσουν. Και επομένω, αυτή η νέα νομοθεσία θα πρέπει να βοηθήσει τις πόλεις κατά την έννοια αυτή. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ζητήσω την Κομισιόν να μας πληροφορεί ε, τακτικά και περιοδικά για τις ε, ε, πράξει τη Επίσης να ζητήσουμε από την Κομισιόν να καλέσει τους εκπροσώπους των πόλεων στις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, στα πιο, στις ε, ε, μεγάλες περιοχές, βεβαίως στις αστικές περιοχές συμφωνώ, αλλά δεν πρέπει να λησμονήσουμε και την Ήπεθρο, γιατί γνωρίζουμε ότι στην Ήπεθρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά και το, το Ταμείο της Γεωργικής Ανάπτυξης, ΦΕΟΚΑ κλπ. Για παράδειγμα, ε, έχουμε επίσης τον μη επιστρεφόμενο ε, ΦΠΑ που σε άλλες περιπτώσεις είναι επιλέξιμος και σε άλλες ε, όχι. Ε, θα πρέπει οι κανόνες να είναι ενοποιημένοι και απλοί. Είμαι πεπισμένος ότι για τις μικρές πόλεις, για τους μικρούς δήμους ε, θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο σημείο επαφής έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν από έναν άνθρωπο, από ένα σημείο όλες τις πληροφορίες που θέλουν και όσον αφορά τα προγράμματα και όσον αφορά ε, τις διαδικασίες πληρωμής. Αυτές δε οι πρέπει να γίνουν όσο γίνεται πιο απλές το σύστημα ε, θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο απλουστευμένο έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν καλά ε, οι πόροι. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει ε, να ταχύνουμε το βήμα μας γιατί ο χρόνος περνάει και δεν θα πρέπει να επιβραδύνουμε την κατάσταση. Ας πάρουμε τις αποφάσεις όσον αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ας μην έχουμε την ίδια καθυστέρηση με το 2007. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάσκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από μακρότατες συζητήσεις αποφάσισε σε ορισμένα μέτρα για την υποστήριξη της υπαίθρου και των νησιωτικών περιοχών αλλά και της ανάπτυξης των αστικών περιοχών, των πόλεων, μικρών και μεγάλων και είναι περιοχές οι οποίες φυσικά παρουσιάζουν πάρα πολλές δυνατότητες στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Είναι διοικητικά κέντρα, είναι οικονομικά κέντρα, είναι κοινωνικά κέντρα και στα πλαίσια της δυναμικής τους, της κοινωνικής την οποία παρουσιάζουν οι πόλεις, αυτές, ε, μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις αλλαγές στις ανάγκες των πληθυσμών που τις κατοικούν. Γι' αυτό θα μπορέσουμε να οργανώσουμε με σωστό τρόπο την προσπάθεια αναδιοργάνωσης και εκ νέου ανάπτυξης του αστικού περιβάλλοντος. Έτσι και μόνο θα καλύψουμε τις ανάγκες των πληθυσμών τους. Βελτίωση της αποδοτικότητας της ενεργειακής των κτηρίων, βελτίωση των ε, μεταφορικών υποδομών, καταπολέμηση της μόλυνσης και σε επίπεδο ατμόσφαιρας και σε επίπεδο ε, θορύβου. Οι ρυθμίσεις αυτές ε, θα ωφελήσουν σχεδόν το 80% του πληθυσμού της Ένωσης εφόσον εφαρμοστούν σωστά. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Αριστερά, Ναυζή, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως κύριε Επιτροπέ, ως μέλος της Διαπραγματευτικής Ομάδας του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι θα θέλαμε οι προσδοκίες που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις αυτές να μπορέσουν να υλοποιηθούν και να βρουν τρόπο χρηματοδότηση στο νέο χρηματοδοτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πρέπει να πούμε όμως ότι δεν είναι πάντα εύκολο να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει η περιφερειακή ε, ανάπτυξη και πολιτική αυτό το ποιοτικό άλμα που χρειάζεται. Το Κοινοβούλιο πάντως θα πρέπει να προχωρήσει ενωμένο και αποφασιστικό. Αλλά η δουλειά που μας περιμένει είναι δύσκολη. Είναι μεγάλη η ανησυχία μου όσον αφορά το επόμενο πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος που ο προϋπολογισμός της πολιτικής συνοχής προτείνεται με μεγάλη μείωση ε, θα πρέπει να κατανοήσουμε το εύρος αυτής της καταστάσεως έτσι ώστε να προσαρμόσουμε την πολιτική μας στο μέλλον αντίστοιχα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, από τους μη εγγεγραμμένους, Στάντλερ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, όλες ε, αυτές ε, οι εκθέσεις έτυχαν τη δική μου υποστήριξη και δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη προσαρμογή των εργαλείων τη πολιτική συνοχή. Και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Επίτροπο που προτίθεται να αναλάβει το έργο αυτό. Ε, επισημάνθηκε από προηγούμενου ομιλητέ η αρχή των συγκοινωνούντων δοκίων. Θα πρέπει να πάψει να ισχύει αυτή η αρχή, γιατί τα κονδύλια τώρα είναι πενιχρά και θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Ε, Ζητούμενο είναι να καταπολεμηθεί βεβαίω η ενεργεία, ιδιαίτερω όταν πρόκειται για τη νέα πολιτική συνοχή στα αστικά κέντρα. Η έκθεση Κοζολίνο ε, προτείνει την ε, θεωρία των κεντρικών τόπων, η οποία έχει αναπτυχθεί εδώ και πολύ καιρό στην αυστρική και γερμανική βιβλιογραφία. Ναι κατά πόσο θα είναι επαρκές να χρησιμοποιηθούν 5% των κονδυλίων για να αναπτυχθούν τα σχετικά εργαλεία δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αρκετό αλλά είναι λογικό να ξεκινήσουμε με νέα εργαλεία και με νέα κονδύλια και στη συνέχεια να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα αυξήσουμε. Ε, δεν, θα είναι και αυτή, δεν θα είναι αυτή η τελευταία προσαρμογή. Τέλος, θα ήθελα να πω, να επισημάνω ένα μεταφραστικό λάθος στο σημείο 10 της γερμανικής μετάφρασης έκθεσης Κοζολίνο όπου ε, τα μέτρα ε, δεν εξυπηρετούν την καταπολέμηση της ενεργειακής αποδοτικότητας αλλά την αύξηση, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Οι υπόλοιποι αγορητέ τώρα θα ξεκινήσουμε με την κυρία Λούκα Τσιγεύσκα για δύο λεπτά. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Polityka spójności jest najważniejszym instrumentem mającym το κλειδί στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η πολιτική συνοχή. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να λιάνουμε κάπως τις περιφερειακές διαφορές και να προχωρήσουμε σε νέες μορφές ανάπτυξης. Ελπίζουμε να ξεφύγουμε από την ύφεση η οποία σώβει σήμερα και θα προσπαθήσουμε τα νέα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε να είναι ευέλικτα και να προσαρμόζονται στις τοπικές ανάγκες. Το ποσοστό θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλό βέβαια γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε σωστά τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Σαν σκιώδη εισηγήτρια έχω πει ότι για να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα στις περιφέρειες μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων θα πρέπει να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος. Θα πρέπει τα πράγματα να είναι πιο απλά, να χρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο έτσι θα πείσουμε και τους πολίτες να δουν με διαφορετικό μάτι και να χρησιμοποιήσουν σωστά τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία πράγματι θα λειτουργήσουν σαν κίνητρο για να απελευθερωθεί το δυναμικό το οποίο κρύβεται πολλές φορές στις τοπικές κοινωνίες. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει επιτέλους μια συζήτηση έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι νομικοί μηχανισμοί, οι τοπικοί συγγνώμη μηχανισμοί που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των κοινοτήτων. Σε στενή συνεργασία με την Ιρλανδική Προεδρία θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλες τους τις περιοχές και τις αστικές περιοχές και τις περιοχές της Υπέθρου μπορούν να αναπτυχθούν εφόσον ληφθούν τα σωστά μέτρα Απαιτούνται λοιπόν σωστές αποφάσεις εκμεταλλευόμενες ακριβώς ε, τις ικανότητες και τις δυνατότητες της κάθε περιοχής ε, μέσω και της σωστής ανταλλαγής εμπειριών και χρηστών πρακτικών ανάμεσα στις χώρες. Ευχαριστώ. Η κυρία, ε, ο κύριος Ολένης Ιγιάκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα θέλαμε να αναφερθούμε σε κάποια βασικά σημεία. Στα με την, ε, σαν με εργαλείο την πολιτική συνοχή θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ένδια. Και υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν ε, να χρησιμοποιηθούν εδώ. Οι πολίτες ε, πρέπει να έχουν δικαίωμα σε παροχή ενέργειας καλής ποιότητας και σε συμφέρουσα τιμή. Και αυτό σε, σε συνδυασμό με την κλιματική πολιτική. Χρειαζόμαστε νέες λύσεις. Άρα χρειαζόμαστε επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό θα αποτελέσει και βάση της ανταγωνιστικότητάς μας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα. Τρίτον, Θέλουμε η πολιτική συνοχή να είναι μια συνολική πολιτική η οποία θα λαμβάνει υπόψη της και τις ανάγκες και τις συνθήκες ε, οι οποίες ισχύουν σε όλες τις περιφέρειες. Ε, και ε, από την άλλη πλευρά βεβαίως θα πρέπει να βοηθήσουμε και τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, μπορούμε να προωθήσουμε ε, είτε το, το αέριο από βιομάζα είτε τη, άλλες μορφές αερίου η που μπορεί να βοηθήσει τους, λιγότε, τους πιο φτωχούς να έχουν πρόσβαση σε ικανή ενέργεια. Πρέπει να βρούμε νέες λύσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάνερ, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ καταρχήν για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Ελέγχθηκατε την ότι η πολιτική συνοχή είναι μια πολιτική με πολλαπλούς στόχους. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε ένα, να εξασφαλίσουμε ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο. Η ενεργική πολιτική είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα είναι όλο και πιο σημαντική στο μέλλον. Γι' αυτό μελλοντικά θα πρέπει να χρηματοδοθεί από το Ταμείο Συνεχή σε ένα μεγαλύτερο τμήμα τη ενεργειακή πολιτική, γιατί είναι αυτή η οποία εξασφαλίζει θέσει εργασία και ανάπτυξη και σε περιφερειακές περιοχές. Η περιφερειακή συνεργασία επίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο εντός της πολιτικής συνοχής, γιατί στο πλαίσιο αυτής της περιφερειακής συνεργασίας μπορούν να αναπτυχθούν βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Και πραγματικά εδώ έχω κάποιε ανησυχίε εν σχέση με την κατεύθυνση που προτείνει το Συμβούλιο για την Περιφερειακή Πολιτική, γιατί μου φαίνεται ότι θέλει να μειώσει τα κονδύλια τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, στην πρόταση Επιτροπής ε, και ε, το Συμβούλιο πραγματικά υπολείπεται κατά πολύ αυτού το οποίο προτείνει το Κοινοβούλιο και ελπίζω η Επιτροπή να πιέσει κάπως περισσότερο το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μιράντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σαν σκιώδης συγγήτρια στον τομέα της ενέργειας θα ήθελα να πω ότι και η πολιτική αυτή θα είναι σε θέση να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την οικολογική αηφόρια. Θα πρέπει να συνδυαστεί λοιπόν με την πολιτική της συνοχής. Πρέπει να έχουμε ε, διαφορές, να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε διαφορές σε σχέση με τους στόχους στον τομέα του περιβάλλοντος. Ξέρουμε ότι εμείς στη χώρα μου σαν παραδείγμα μπορούμε να εξάγουμε ενέργεια στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρήζει μερικές φορές διορθώσεων βέβαια γιατί η ενέργεια πολλές φορές μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις από τον τόπο παραγωγής της με ό,τι αυτό σημαίνει θα πρέπει να προωθήσουμε και άλλες πηγές ενέργειας, εναλλακτικέ πηγές οι οποίες να διαμορφώνουν σωστές τιμές και όχι υπερβολικές τιμές. Το σημείο 12 της έκθεσης δεν είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, ξεκάθαρο για τις λεγόμενες διεθνικές ή προσωρινές πηγές ενέργειας. Τι ακριβώς εννοεί Μίκολσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους εισηγήτες του Κοινοβουλίου και τις διαπραγματευτικές ομάδες για ένα καλό πακέτο στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Δεν θα τεθεί σε λειτουργία βέβαια το 13 ή 14, αλλά όταν τα πράγματα οριμάσουν. Αυτή η νέα κατηγορία των λεγόμενων μεταβατικών περιοχών θα περιλαμβάνει και τη δική μου περιφέρεια της Βόρειας Ιρλανδίας. Θα πρέπει να στηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κατηγορία αυτή θα παίξει ένα σημαντικότατο ρόλο παράλληλα με την λεγόμενη ειρηνευτική χρηματοδότηση την οποία έχουμε εδώ και αρκετό καιρό και που έχει συνεισφέρει τα μάλα στην Βόρεια Ιρλανδία τα τελευταία χρόνια. Η συνέχεια του Ταμείου Ειρήνευσης είναι καθοριστική για το μέλλον βέβαια της χώρας μου, της περιοχής μου μάλλον. Θα ήθελα λοιπόν να μας διαβεβαιώσατε ότι η πρόταση η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο ε, για, τον, ε, για τη συνέχιση του προγράμματος αποκατάστασης της ειρήνης ε, θα συνεχιστεί. Πρέπει όμως να ξεκαθαριστεί ποιοι θα το χρηματοδοτήσουν, ποια θα είναι η πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι επιπλέον χρήματα όπως στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει να είναι φετούλες και κομματάκια από το Περιφερειακό Ταμείο ή από το Ταμείο Συνοχής που έτσι και αλλιώ κάνουν εξαιρετική δουλειά στα σύνορα της περιοχής μου και θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν. Θα πρέπει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες και να καταλήξουμε στις σωστές αποφάσεις. Και εμείς στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να πάρουμε τις σωστές κατά προτεραιότητα αποφάσεις για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω για το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο επανειλημμένα έχει χρησιμοποιηθεί από τη χώρα μου. Υπενθυμίζω ας πούμε το σεισμό στην Ούμπρια, αλλά και πιο πρόσφατα ε, στην τραγωδία που έλαβε χώρα στην ε, Εμίλια Ρωμάνια. Ε, και τα προβλήματα τα οποία προκάλεσε στο Βένετο ε, η μεγάλη πλημμύρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ταμείο, αλλά ε, έχει και όρια. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τα χρονικά περιθώρια. Μια βοήθεια που φτάνει αργά είναι σχεδόν ανώφελη. Θα πρέπει σε περίπτωση καταστροφής να μπορούν άμεσα να χρησιμοποιηθούν τα μέσα τα σωστικά και με μεγάλη ευελιξία και στην περίπτωση του ε, Βένετο ε, που υπέστη καταστροφές από πλημμύρες περιμένανε σχεδόν ένα χρόνο μέχρι να φτάσει η βοήθεια ε, λόγω των γραφειοκρατικών προβλημάτων. Εδώ και δύο χρόνια ξανασυζητάμε τον κανονισμό που ε, διέπει το Ταμείο αυτό. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ξαναγράψουμε τους κανόνες ε, αυτού του ε, οργάνου έτσι ώστε να μπορεί να βοηθήσει πραγματικά σε περιπτώσεις ζημιών, σε περιπτώσεις καταστροφών γιατί διαφορετικά τα θύματα είναι αυτά τα οποία θα πληρώσουν για μία ακόμα φορά. Θα πρέπει να κατεβεί το ελάχιστο κατόφλι. Θα πρέπει να πάρουμε ε, υπόψη μας και το γεγονός ότι την επόμενη δεκαετία σίγουρα θα αυξηθεί ο ρυθμός και η πυκνότητα αυτών των μεγάλων ε, καταστροφών. Ε, βλέπουμε ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές. Θα πρέπει η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο στην πρόληψη έτσι ώστε να αποφύγει τουλάχιστον τις τραγωδίες οι οποίες μπορούν να αποφευχθούν. Ευχαριστώ. Η κυρία Έρνστε για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι πραγματικά μια ξεκάθαρη ενίσχυση της αστικής διάστασης, διάστασης των πόλεων, γιατί οι πόλεις είναι πολύ σημαντικές όσον αφορά τι δημογραφικές ε, μεταβολές αλλά και την κοινωνική ανισότητα. Και δεν θα πρέπει να περισσορίσουμε σε μεγαλόσχημα λόγια, αλλά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν μια μείζωνα πρόκληση των καιρών μας και αντιστοίχως θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις προτάσεις. Και εδώ πραγματικά έχω κάποιες ε, ανησυχίες όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι πόλεις έχουν μια ιδιαίτερη σημασία για την ύπεθρο που τις περιβάλλει και είναι τόποι δημογραφικής ανάπτυξης. Από τη μία έχουμε ε, ε, φαινόμενα αστιφιλίας αλλά και εξόδου από τις ε, πόλεις. Οι Ρωμά εκδιώκονται από τις πόλεις. Το στίγμα της φτώχειας διαρριγνύει τον αστικό ιστό. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν καθόλου περικοπές στον τομέα αυτό της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μόλτσερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το πόσο σημαντική είναι σε μια περίοδο κρίσης μια μακροπρόθεσμη χάραξη στόχων ε, μας δείχνει το παράδειγμα της φούσκας των ακινήτων που έσκασε στην Ισπανία. Βλέπουμε ότι στο, στο ζήτημα της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης ε, το, η περίοδος ε, ε, απόσβεσης είναι πολύ υπερβολικά μεγάλη λόγω της ε, αλλαγής του πολιτικού πλαισίου θα πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο την πολιτική μας προς συγκεκριμένους στόχους. Θα πρέπει να υπάρξει ε, μεγαλύτερη, περισσότερη ποιότητα, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν πιο εύχριστα αποτελέσματα μιας πολιτικής η οποία επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους στόχους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βανίστερο για δύο λεπτά. Ε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή η συζήτηση στην ε, Ολομέλεια ε, μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε σε βάθος πράγματα τα οποία έχουμε ε, ήδη συζητήσει και στο παρελθόν ε, και οι χώρες επίσης έχουν συζητήσει τέτοιου είδους θέματα με την Κομισιόν και όταν μιλούν για ενέργεια και για, όταν μιλάνε για αστική ανάπτυξη. Βεβαίως θα πρέπει οι κανόνες να αλλάξουν, θα πρέπει να προχωρήσουμε με άλλο τρόπο. Μιλάμε τώρα για το Ταμείο Αλληλεγγύης, μιλάμε για βοήθεια που θα πρέπει να δοθεί και να δίνεται σε περιπτώσεις ε, ε, φυσικών ή άλλων καταστροφών. Αλλά τώρα ε, θα πρέπει να δοθούν οι δυνατότητες να γίνουν επενδύσεις για πιο ευφυή, για πιο πράσινη, για πιο καινοτόμα Ευρώπη. Πιστεύω ότι αυτή η ευφυής εξειδίκευση είναι κάτι που χρειαζόμαστε ε, το χρειαζόμαστε αυτήν την ε, ευφυΐα έτσι ώστε να έχουμε την πραγματική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα πρέπει να επιταχύνει το ρυθμό της ε, η Ευρώπη γιατί μέχρι τώρα πολλές επικαλύψεις έχουν υπάρξει. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει στο μέλλον. Θα πρέπει να γίνεται καλύτερα η δουλειά μέσω και της συζήτησης που κάνουμε τώρα θα πρέπει να δούμε εάν ε, ε, πραγματικά και τα κράτη-μέλη ακολουθούν ε, στις επαφές που έχω με τις, στις διάφορες χώρες μέλη καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλές δυνατότητες το δυναμικό είναι εκεί οι πρωτοβουλίε είναι εκεί αλλά δεν υπάρχει αρκετή επικοινωνία μεταξύ των χωρών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά το Ταμείο Συνοχής να αποκτήσει πραγματικά πραγματική, πραγματικό περιεχόμενο πριν τις ε, χριστουγεννιάτικες ε, εκλογές, ε, συγγνώμη διακοπές, είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση αυτή. Πρέπει να την ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Σταυρακάκης. Παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης και την πολύ καλή έκθεσή της θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ενώσω τη φωνή μου με, όλου με υποστηρίζουν ότι το ταμείο αλληλεγγύη αποτελεί ένα από τα κύρια και πιο επιτυχημένα μέσα έκφραση αλληλεγγύη που διαθέτει η ευρωπαϊκή ένωση. τα τελευταία χρόνια έχει επανειλημμένω γίνει κινητοποίηση του ταμείου για αρρωγή σε πληγέντα από καταστροφές κράτη μέλη. ωστόσο έχουν διαπιστωθεί ορισμένα προβλήματα στη διαδικασία κινητοποίηση και εφαρμογή του με συνέπεια οι διαθέσιμοι πόροι να καθυστερούν να φτάνουν στι περιοχέ μια καθυστέρηση που δημιουργεί προβλήματα στην παροχή βοήθεια τη στιγμή που η βοήθεια αυτή είναι πιο αναγκαία από οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή. γι' αυτό το λόγο η σοσιαλιστική μα ομάδα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο υποστηρίζει ένα πιο ευέλικτο αποτελεσματικό και πλουστευμένο ταμείο εύκολο και γρήγορο στην κινητοποίησή του το οποίο επιτρέπει στην ευρωπαϊκή ένωση να ανταποκριθεί καλύτερα στι σοβαρέ καταστροφέ παρέχοντα έγκυρη ανακούφιση για του πολίτε που την έχουν ανάγκη αυτή οφείλει να είναι η ουσία της αλληλεγγύης που προσφέρει η ένωσή μας στους πολίτες της. Ευχαριστούμε πολύ. Ως επόμενος ομιλητής έχει το λόγο για ένα λεπτό ο κύριος Βαντάλεν. Helaas is het zo dat er eh, regelmatig berichten opduiken over onjuist gebruik van subsidies uit de cohesie en structuurfondsen. Έχουμε πολύ συχνά εκθέσεις για αναποτελεσματική χρήση των πόρων του Ταμείου Συνεχής. Όπως έγινε για παράδειγμα στην Πολωνία που τα χρήματα κατέληξαν ε, στα χέρια των πολυεθνικών. Στην ε, Πολωνία ε, βάλαμε κάποιους υγιείς φραγμούς για την χορύπανση αλλά κανείς δεν φαίνεται να ενοχλείται. Νομίζω ότι θα πρέπει επίση με χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωσης να χρησιμοποιηθούν δρόμοι για μοτοποδήλατα στην Ολλανδία. Έχει αυτό κανένα νόημα. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι τα κονδύλια από τα τομεία πραγματικά να εισραίουν προ τι φτωχέ περιοχές. Αυτό είναι το νόημα. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια υπεραξία σε τοπικό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος για τη χρήση των ε, χρημάτων μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επαρκείς αιτιολογήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ως επόμενο ομιλητή για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριο Τσιμάνσκι. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούμε όλοι για να πούμε ότι η πολιτική συνοχή έχει θετικέ επιπτώσει στην οικονομική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε κάποιες περικοπές που έγιναν στο συγκεκριμένο τμήμα του προϋπολογισμού. Οι περικοπές αυτές είναι απολύτως λανθασμένες. Θα πρέπει να ενθυμούμεθα επίσης ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να δαπανηθούν με τον σωστό τρόπο. Αν η λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνει δεκτή, τότε κατά τη διάρκεια της επομένης δημοσιονομικής περίοδου τα μισά οι μισές πιστώσεις από το Περιφερειακό Ταμείο θα στραφούν αποκλειστικά στο θέμα των δραστηριοτήτων ε, για την προστασία από τις κλιματολογικές αλλαγές. Αυτό δεν είναι ο σωστός τρόπος για να προχωρήσει η οικονομία μας. Για κάποιες χώρες σαν τη δική μου, οι οποίες βασίζονται δυστυχώς ακόμα στον άνθρακα, αυτό θα είναι καταστροφή, το να ξοδεύουμε το 50% των χρημάτων τα οποία μας δίδονται για την ε, οικολογική πλευρά αν θέλετε της αντιμετώπισης του προβλημάτων. Ε, υπάρχουν δυνατότητες που οποίες θα πρέπει να εξετάσουμε όπως ε, το φυσικό αέριο από λίθους και τα λοιπά είναι θέματα τα οποία είναι από ό,τι φαίνεται ε, μορφές παραγωγής καθαρότερες από την παραγωγή από πετρέλαιο και έτσι θα αποφύγουμε τους κινδύνους τους οποίους έχουμε μπροστά μας όταν συζητήσουμε εκ νέου το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Τώρα για το Ταμείο Αλληλεγγύης θα πρέπει να υποστηρίξουμε την εισηγήτρια όταν ζητά την παράταση και το streamlining αυτού του συγκεκριμένου μέσου η συγγήτρια πάρα πολύ σωστά λέει ότι είναι ένα από τα πολύ λίγα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να επιδείξουμε την αλληλεγγύη μας προς τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Και εδώ θα συμφωνήσω ειδικά με τον κύριο Βαντάλεν ε, για το ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη, ή περισσότερο ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητή για ένα λεπτό, κύριο Σαγκουράκη. Ο κοινό τόπο και των τριών εκθέσεων είναι η διάθεση δημοσίου χρήματο στου μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου προκειμένου να κινητοποιήσουν τα συσσωρευμένα κεφάλαιά του και να ξεπεράσουν την καπιταλιστική κρίση σε βάρο των εργαζομένων. Συγκεκριμένα καλούν την τοπική διοίκηση να συνάψει εταιρικέ σχέσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα καθορίζουν την επιλεξιμότητα των έργων και τον τρόπο διάθεση του των κονδυλίων όχι για την ικανοποίηση των οξυμένων λαϊκών αναγκών που είναι ιδιαίτερα ε, σήμερα μεγάλες όπως οι δημόσιες δωρεάν συγκοινωνίες αντισυσμική και αντιπλημμυρική προστασία υποδομές δημόσιας εκπαίδευσης και υγείας κτλ. αλλά αντίθετα σε νέους κερδοφόρους τομείς για το κεφάλαιο όπως η διαχείριση απορριμμάτων εμπορική εκμετάλλευση ιστορικών και πολιτισμικών μνημείων απελευθέρωση της παραγωγής και διανομής ενέργεια οι εκθέσει προωθούν την αντιλαϊκή στρατηγική ευρώπη 2020 που απορροφά ήδη το 63% των κοινοτικών πόρων στην ελλάδα. 40% των πόρων επιστρέφει απευθεία στους μεγάλου μονοπωλιακού ομίλου και το υπόλοιπο 60% πάει στην ελληνική ολιγαρχία για, να εντείνει τι καπιταλιστικέ αναδιαρθρώσεις. Η όξυση των γεωγραφικών και κοινωνικών αντιθέσεων στο καπιταλιστικό σύστημα αποτελεί νομοτέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενο ομιλητή είναι ο κύριος ε, Τσέλερ. Για λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι καλό ότι ε, εν ώψη της, ε, των συνεχιζόμενων τριμερών συνομιλιών φαίνεται από τις εκθέσεις πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της πολιτικής συνοχής. Είμαι ιδιαίτερο ευγνώμων για την έκθεση του συναδέλφου Κοζολίνου, ο οποίο πολύ γλαφυρά μα έδειξε πόσο σημαντικά είναι τα θέματα τη ανάπτυξη των πόλεων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εγώ ε, είμαι. Ε, ο κ. Χάν είπε ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής μπορούν να επιτευχθούν μόνο εφόσον εφαρμοστούν στους αστικούς ε, χώρους όπου ζουν το 70% του ευρωπαϊκού ε, πληθυσμού και όπου υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη. Ε, και έχει λεχθεί κατά επανάληψη πόσο σημαντική είναι η βιώσιμη ανάπτυξη στην διακήρυξη του Μπρίστολ αλλά και του Τολέδο διακηρύσσονται αυτοί οι στόχοι. Ε, έχει έρθει η ώρα να γίνουν ε, πράξη αυτές οι υποσχέσεις και οι πόλεις να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα διορθωτικά ταμεία και να πάρουν τη θέση που τους ανήκει στις, ε, συμφωνίες, στις εταιρικές συμφωνίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ως επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, ο κύριος Νίλσον. Παρακαλώ. Eh, Συνάδελφοι, για το ποιο είναι ο ρόλο τον οποίο θα πρέπει να παίξει η πολιτική συνοχή, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε σαφείς. Μπορεί να παίξει ένα σημαντικότατο ρόλο και σε ορισμένε περιφέρειες αποφασιστικότατο ρόλο. Η εμπειρία μου ε, βασίζεται στη Βόρεια Σουηδία. Πριν 6 χρόνια δημιουργήσαμε το περιφερειακό πρόγραμμα και αποφασίσαμε να κινητοποιήσουμε κυρίως την ανάπτυξη λύσεων ε, εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Οδηγηθήκαμε λοιπόν σε μια έκρηξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασχολούνται με την τεχνολογία και με την εξοικονόμηση ενέργειας. δημιουργήθηκε ένας πολύ σημαντικός αριθμός θέσεων απασχόλησης με αυτόν τον τρόπο. Υπήρξε καινοτομία σημαντική και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και η εξοικονόμηση ενέργειας στην δασοκομεία σαν παράδειγμα μας ανοίγει το δρόμο και για εξοικονομήσεις σε άλλους τομείς. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομιλήτρια για ένα λεπτό η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σε αυτούς τους ε, χαλεπούς ε, οικονομικούς καιρούς ε, θα πρέπει να γινόμαστε φιέστεροι έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Θα πρέπει οπωσδήποτε όμως να κινηθούμε και βάσει της στρατηγικής και των στόχων του 2020. Καλωσορίζω λοιπόν την εργασία των εισηγητών. Κυρίως στηρίζω τον ρόλο που πρέπει να παίξει η επικουρικότητα. Επίσης χαίρομαι γιατί βλέπω ότι γίνεται έτσι μια προσπάθεια ε, ε, ευελιξίας. Όλα αυτά, εάν συνδυαστούν με την έμφαση που πρέπει να δοθεί στην θεματική συγκέντρωση ε, για περιοχές όπως ας πούμε η Ουαλία, σίγουρα θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα και θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό των διευθυντικών ταμείων. Όμως, γιατί λυπούμε, αλλά υπάρχει πάντα ένα όμως. Ε, θα πρέπει να υπάρξουν οι απαραίτητες διασφαλίσεις. Θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν οι απαραίτητες διασφαλίσεις έτσι ώστε πραγματικά αυτοί που χρειάζονται τα χρήματα περισσότερο να τα λαμβάνουν. Αλλά βλέπουμε ότι αυτές αποσιάζουν. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής ε, για ένα λεπτό, κύριος Μάτουλα. Η πολιτική συνοχής είναι ένα επενδυτικό μέσο το οποίο αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και εξασφαλίζει θέσεις εργασίες. Ε, οι περικοπές στο πεδίο της πολιτικής συνοχής, ε, στο πλαίσιο του MFF, ε, θα μειώσουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και θα μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι. Οι στόχοι. Και επίσης οι περιφερειέ τη σύγκληση θα πληγούν ανεπανόρθωτα. Η εδαφική συνεργασία είναι ένα σημαντικός παράγον για την μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των ε, περιφερειών στην Ευρώπη και εδώ θα υπάρξουν σημαντικέ επιστοχωρήσει. Οι αστικέ περιοχέ βεβαίω είναι ιδιαίτερω σημαντικέ και έχουν ένα ρόλο κλειδί. Γι' αυτέ η ανταγωνιστικότητα είναι ιδιαίτερο σημαντική γιατί είναι ο βασικό κινητήρα για την εξασφάλιση θέσεων απασχόληση. Γι' αυτό η μετανάστευση προς τις πόλεις αυξάνεται, η αστιφιλία αυξάνεται και στην Ευρώπη. Οι πόλεις ωστόσο είναι αυτές που εκτίθενται περισσότερο στην κρίση και στα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης. Αυτό έχει ολέθριες κοινωνικές πεπτώσεις και βλέπουμε παιδιά να υποφέρουν, έχουμε φαινόμενα αποκλεισμού, ακόμα και η κλιματική μεταβολή είναι εδώ σημαντική. Θα πρέπει να έχουμε ταχύες αντιδράσεις και να ανταπεξέλθουμε στις τοπικές ανάγκες. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αυξήσει τις διοικητικές ικανότητες στις πόλεις, θα πρέπει οι οικονομικοί παράγοντες να ενισχυθούν μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων και να ενισχυθούν τα αστικά δίκτυα. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομιλήτρια για ένα λεπτό, η κυρία Ιριγκοβέν Πέρες. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Πράγματι η περίοδο κρίσης στην οποία βιώνουμε περιπλέκει τις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας αλληλέγγυας Ευρώπης. Πρέπει σε δύσκολους καιρούς να βρούμε λύσεις όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές πλευρές της ύφεση, αλλά και να αποφύγουμε μια κοινωνική διάλυση γιατί η πολιτική συνοχή έχει δείξει μέχρι τώρα πόσο αποτελεσματική είναι σε επίπεδο συνεκτικό και ανταγωνιστικό. Θέλω να συγχαρώ εδώ τους συζητητές τίνουν επίσης το να ζητήσουν την κοινωνική αηφορία και την ανανέωση των αστικών περιοχών. Πρέπει να ζητήσουμε μια αποτελεσματική και ευέλικτη και εύκολα προσαρμοζόμενη πολιτική συνοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει εμείς να ακυρώσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής αυτής ιδιαίτερα στις περιοχές και τις χώρες που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφε. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος ε, Μπίλαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σε σχέση με την έκθεση της κυρίας Κολάρτσα Μπομπίνσκα, ε, θεωρούμε ότι ε, πραγματικά ένας μεγάλος στόχος που έχουμε είναι η διασφάλιση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενεργειακή μας πολιτική να ελέγχουμε τις εισαγωγές και από την άλλη πλευρά να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις, τους τοπικούς τις τοπικές δυνατότητες παραγωγής ενέργειας, να χρησιμοποιήσουμε νέες μορφές όπως είναι το σχιστολιθικό αέριο, ε, βεβαίως θα πρέπει να ε, μπορέσουμε να βοηθήσουμε οικονομικά ε, και τις περιοχές αυτές οι οποίες ούτε δυνατότητα τοπικής παραγωγής ενέργειας έχουν αλλά και έχουν πληγεί ιδιαίτερος από την κρίση. Καλή ενεργειακή συνεργασία με χώρες εταίρους που είναι όμορες κυρίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε επενδύσει αρκετά ε, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά τα ορυκτά παραμένουν πρώτα στη σειρά. Ευχαριστώ, πολύ. Λυπούμε που πέρασε ο χρόνος σας. Ε, επόμενη μιλήτρια είναι η κυρία Σάντσεθ Σμιτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές οι τέσσερις εκθέσεις όλες βασίζονται στην αρχή της οικονομικής αλληλεγγύης μεταξύ ε, των εδαφών. Και ε, το Ταμείο Ελεγγύης έχει ήδη δώσει πολλά εκατομμύρια ευρώ στις χώρες ε, μέλη ε, από το 2002 στις ε, περιπτώσεις 49 φυσικών καταστροφών. Ωστόσο, παρόλα αυτά, οι προθεσμίες είναι υπερβολικά μεγάλες, οι διαδικασίες πολύπλοκες, τα, η γραφειοκρατία επαχθείς και οδηγούν σε, σε πολλές απογοητεύσεις στους πολίτες. Τα θέματα που αναφέρονται στις τρεις άλλες εκθέσεις, ε, ε, μηχανισμός συντονισμός των ταμείων, ε, ε, επιπτώσεις ενεργειακή πολιτικής κλπ. Είναι η ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί ε, στα θέματα αυτά μελλοντικά. Ε, πρόκειται για μια θαυμάσια επένδυση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Επιτρέπει προγράμματα κοινωνικής συνοχής στις πόλεις, την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια, την ε, διαφύλαξη των φυσικών πόρων κλπ. Στην τελευταία πρόταση, ε, πρόταση για τον προπολογισμό, ε, ε, προβλέπεται 27% εδαφικής συνοχής. Θα πρέπει ωστόσο ο προϋπολογισμός να είναι επαρκής για να υπάρξουν ορατές, ορατά αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφε. Ο κύριος Διάντζελης έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πολιτική συνοχή είναι πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη, για την εργασία. Η καλή χρήση αυτών των πόρων είναι απαραίτητη. Είμαι ικανοποιημένος από την εργασία που βλέπω, γιατί βλέπω ότι γίνονται σημαντικά βήματα προς τα εμπρός, έτσι ώστε να ε, ε, έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών αρχών ε, στην διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η σωστή χρήση και ολοκληρωμένη χρήση ε, των ε, ευρωπαϊκών πόρων έτσι ώστε σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς να επιλεγεί ο η μορφή αυτή η οποία ε, είναι πιο σωστή ε, και η ε, δοκούσα για τις τοπικές ανάγκες. Θα πρέπει να συνεργαστούν λοιπόν σε ένα ευρύ φάσμα οι πρωταγωνιστές και οι ενδιαφερόμενοι με στόχο βεβαίως πάντα να γίνει πιο κοντινή μικρή απόσταση ανάμεσα στον πολίτη και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Τειξέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση αυτή η οποία γίνεται σήμερα σύντομα σχετικά μετά από τη στιγμή που η Πορτογαλία ζήτησε από την Επιτροπή την κινητοποίηση του συγκεκριμένου ταμείου λόγω των προβλημάτων των καιρικών συνθήκων των προβληματικών τον προηγούμενο Δεκέμβριο. τα στάδια γενικά τα οποία ακολουθούνται για την κινητοποίηση ε, του Ταμείου Αλληλεγγύης ε, είναι μερικές φορές ε, δύσκολα και μακροχρόνια. Υπάρχουν καταρχάς κάποιες αντιφάσεις ανάμεσα στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση φυσικών καταστροφών θα μπορούσε να είναι σε θέση να αντιδράσει έγκαιρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά όχι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση της Μαδέρας χρειάστηκαν κύριοι δύο χρόνια για να φτάσει η βοήθεια. Αυτή είναι η κατάσταση της άμεσης ανταπόκρισης στους πληθυσμούς που έχουν φυγεί. Θα πρέπει λοιπόν και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αλλά κυρίως το Συμβούλιο το οποίο έχει μπλοκάρει τη δράση μέχρι τώρα να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του συστήματος ή να πει ότι εντάξει η λέξη αλληλεγγύη νόημα πια δεν έχει γιατί εκφράζεται πάντα με τέτοια καθυστέρηση. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, κύριο Σταμπάντη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βόν για την έκθεσή του γιατί τονίζει το σημαντικό στόχο της πολιτικής συνοχής που είναι ακριβώς η συνοχή των φτωχών ε, περιοχών. Είναι απαράδεκτο ε, να μειώνονται τα κονδύλια που δίδονται στις φτωχές περιοχές. Από το 2014 ε, θα πρέπει να ληφθούν εντονότερα υπόψη οι φτωχότερες περιοχές. Από τις 7 περιοχές της Ουγγαρίας, 6 βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση φτώχες. Γι' αυτό είναι, απαράδεκτο, ε, είναι απαράδεκτο συγγνώμη, να μειωθούν τα κονδύλια που θα λάβει η Ουγγαρία προσεχώς κατά 30%. Θα ήθελα να παρακλέσω τον Επίτροπο κύριο Χάν να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση για αυτό το πρόβλημα. Και θα πρέπει να μεριμνήσουμε ούτως ώστε οι, κανόνες να μην ε, καθιστούν ε, αδύνατο να χορηγούνται αυτά τα χρήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Μάζεχ Κούκοβιτς. Κύριε Επιτροπέ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης ε, είναι απαραίτητο αλλά στο μέλλον χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Τα κριτήρια θα πρέπει να απλουστευθούν ε, και θα πρέπει η κοινοποίηση των στόχων να είναι ε, πιο σαφής. Ε, ξέρουμε ότι στις φυσικές καταστροφές ιδιαίτερα όποιος ανταποκριθεί πιο γρήγορα είναι σαν να δίνει τα διπλά, σαν να προσφέρει τα διπλά. Ε, στις φυσικές καταστροφές λοιπόν μπορούμε να αποφύγουμε ε, πάρα πολύ μεγάλες περαιτέρω επιπτώσεις. Ε, ξέρουμε ότι όσον αφορά την ενέργεια τώρα ότι υπάρχουν πολλοί αναξιοπαθούντες πολίτες οι οποίοι λόγω της κρίσης έχουν μείνει χωρίς τίποτα. Η γεωγραφική θέση της Σλοβενίας είναι ένα ακόμα περισσότερο αρνητικό στοιχείο που επιδεινώνει την ε, κατάσταση. Η Σλοβενία έχει ζητήσει βοήθεια, έχουμε ετοιμάσει ψήφισμα και ζητώ να το στηρίξετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Βεστφάλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι η πολιτική των πόλεων είναι η πολιτική του μέλλοντος, γιατί οι πόλεις είναι κινητήριες δυνάμεις ε, μιας βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Ε, ένα πολύ μεγάλο ποστό του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ παράγεται στις πόλεις. Ταυτόχρονα θα πρέπει ωστόσο να αναγνωρίσουμε ότι η αστικοποίηση έχει και μια ε, ζωφερή πλευρά. Οι πόλεις ε, πάσχουν από ρήπανση, πεπαλαιωμένες δομές και από τις δημογραφικές μεταβολές. Γι' αυτό η Ευρώπη χρειάζεται μια φιλόδοξη πολιτική για τις πόλεις. Η έκθεση του συναδέλφου Καζολίνο κατά την άποψή μου φωτίζει μια σημαντική πτυχή, δηλαδή το πώς ε, μπορεί η εξηγένση των πόλεων τελικά να εξασφαλίσει μια οικονομική ανάπακαμψη. Ε, το ΕΦΡΕ ε, παίζει σημαντικό ρόλο και σχετικές διαπραγματεύσεις προσπαθούμε να πετύχουμε κάποιες βελτιώσεις ώστε να έχουμε μια βιώσιμη και η οικολογική εξυγένση των πόλεων. Γιατί αυτό ακριβώς χρειάζονται οι πολίτες ως αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής των πόλεων. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Και τώρα ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των επίσημων ομιλητών και τώρα θα έρθουμε στη διαδικασία Catch the Eye και έχω τον άχαρο ρόλο γιατί πραγματικά βρισκόμαστε σε μεγάλη χρονική καθυστέρηση από τον προηγούμενο πρόεδρο ε, και από την άλλη υπάρχουν ε, πάρα πολλοί ε, που ζήτησαν το λόγο να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία του Catch the Eye. Θα πρέπει να κάνουμε ένα επιμερισμό βάσει του φίλου και της πολιτικής ομάδας. Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Μπάνκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή η οποία ασχολείται με τα αστικά κέντρα είναι σημαντικό στοιχείο της πολιτικής συνοχής. Εδώ στο σημείο 4 θα πρέπει να ενεργοποιηθούν συγκεκριμένοι πόροι ούτω ώστε οι εξόχω απόκεντρε ε, ε, περιοχέ να μπορέσουν να σωματωθούν στην κοινωνία. Στο σημείο 7 αναφέρεται ότι χρειαζόμαστε νέες ε, μορφές της εξυγίανσης των πόλεων. Γιατί εδώ θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε κάποιες αθλητικές δραστηριότητες εντός της ψυχαγωγίας των ε, πολιτών. Ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική ένταξη ο αθλητισμός δίνει και στα παιδιά μας μια δυνατότητα να ζήσουν χωρίς ναρκωτικά και αλκοόλ. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε παιδικές χαρές όπου να μπορούν να παίζουν τα παιδιά μας. Και επίσης χρειαζόμαστε μια παιδαγωγική, μια εποπτεία των παιδιών. Στην ε, Ουγγαρία υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Γιόρνταν για ένα λεπτό. Θα πω δύο λόγια όσον αφορά την έκθεση της συναδέλφου Κολάσκα Μπομπίνσκα. Πρόκειται για εξαίρετη έκθεση και θέλω να τη συγχαρώ τη συνάδελφο. Η ενεργειακή πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχει μεγάλες επιπτώσεις και στην οικονομία στο σύνολό της, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και βεβαίως και στην παραγωγή το ε, μόλυνσης διοξιδίου ε, του άνθρακος. Η αηφόρος ε, ενέργεια, οι αηφόρες μορφές ενέργειας κοστίζουν περισσότερο. Ε, αυτό είναι αλήθεια και επενδύσεις μπορούν να γίνουν κατά αυτή την έννοια, μονάχα έννοια η οικονομία είναι δυνατή. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε το Ταμείο Συνοχής ε, και θα πρέπει όλες οι χώρες να συνδράμουν έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει σε αυτούς όσον αφορά την ενέργεια και όσον αφορά και το περιβάλλον. Ε, θα πρέπει να δούμε ευφιέστερους τρόπους πρόθεση της ενέργειας ε, και για οικιακή χρήση και όσον αφορά την ε, διακρατική, τις διακρατικές συμφωνίες. Ευχαριστώ. Mrs. Jordan, would you accept a blue card from Mrs. Δέχεστε από την κυρία Τικάου μία μπλε κάρτα. Please. întreb pe doamna Jordan dacă consideră că doar energiile... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μάθω εάν πιστεύει ότι μόνο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυτές που θα πρέπει να προωθηθούν. Ή μήπως θεωρεί ότι τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί μέχρι σήμερα για την ενεργειακή αποδοτικότητα των λεγόμενων των κατοικιών μάλλον ε, είναι ανεπαρκή νομίζω ότι έχουμε ανάγκη τουλάχιστον 10 με 15% για να διασφαλίσουμε και τις σωστές, ε, τα σωστά αποτελέσματα στις πόλεις. Eh, Δεν είμαι βεβαία ότι σας κατάλαβα καλά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ε, στις ε, επόμενες, στο επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο έχουμε υπογραμμίσει ε, την ανάγκη για χρήση ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στο επόμενο θα θελήσουμε, το σωστό είναι, να ε, εφαρμοστούν καλύτερα όλοι αυτοί οι κανόνες οι οποίοι αφορούν ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια στα σπίτια. Ναι, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. κυρία Ζηνιαλόβα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Η εδαφική συνοχή είναι μία από τις βασικές αρχές της στρατηγικής 2020. Θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει συνεπώς να υποστηρίξουμε αυτές τις ε, φτωχές ε, περιοχές στις διαπραγματεύσεις εγώ ήμουν ε, εισηγητής για την Επιτροπή Μεταφορών και έδωσα, τόνισα ακριβώς αυτό το σημείο, δηλαδή ότι είναι σημαντική η εδαφική συνοχή και η ανάπτυξη των υποδομών στις φτωχότερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από το 2000 στο 2020. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο τα κονδύλια τα οποία προορίζονται για τις ε, περιοχές, συνοχές, ε, περιοχές συνοχής να μειώνονται. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές θα πρέπει κατά την άποψή μου να έχουν μια πιθανότητα να προετοιμάσουν ποιοτικά προγράμματα και να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κονδύλια που τους δίδονται. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Άλβες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ η διασυνοριακή συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Μιλάμε βέβαια και για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Αζόρες, ας πούμε, ε, βρίσκονται στον Ατλαντικό ε, ανάμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ε, η Αζωριανή Διασπορά είναι τετραπλάσια από τους κατοίκους των ε, Αζωρών, δηλαδή αυτοί που ζουν δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθούν όλες οι ευκαιρίες για αυτούς που εξακολουθούν και μένουν στα νησιά αυτά αλλά ε, να ε, μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και την βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών έτσι ώστε ε, να αυξηθεί ο βαθμός καλής διαβίωσης των κατοίκων των Αζωρών. Ναι, μια καλή συνεργασία λοιπόν με τους εταίρους, έστω και αν δεν είναι όμοροι οι γείτονες αυτοί. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φερέιρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι δυνατόν σε μια κοινή συζήτηση ε, να μπαίνουν ε, θέματα ε, τα οποία από μόνα τους θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο μεγάλης ε, συζήτησης. Ε, ο ρόλος τη πολιτικής συνοχής, α πούμε, θα έπρεπε να συζητηθεί από μόνο του. Γνωρίζουμε ότι η χρόνια έλλειψη μέσων και εργαλείων ενισχύθηκε από την παρούσα κρίση δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε χωρίς να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τα εργαλεία στα πλαίσια μιας εμβάθυνσης της ολοκλήρωσης ε, γιατί διαφορετικά ε, θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό πραγματικά. Ε, έγινε λόγος για ανάγκη διπλασιασμού του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού κάναμε ένα σωρό διευρύνσεις και όχι μόνο δεν αυξήθηκε ο προϋπολογισμός αλλά το βαίνει μειούμενος και τώρα θέλουν να τον μειώσουν ακόμα περισσότερο. Μα τότε θα αρχίσουν να υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες αποκλήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε συνάδελφε. Ε, τελευταίος ομιλητής στη δικασία Κάτσου Διάη, ο κύριος Όμπερ Μάιερ για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ε, έχει νόημα πράγματι να γίνει μια πιο επακεντρωμένη εφαρμογή της στρατηγικής, δηλαδή να συμμετάσχουν οι τοπικοί ε, φορείς. Ωστόσο θα πρέπει εδώ να είμαστε προσεκτικοί γιατί ε, το ξέρουμε και από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, ε, στα σημεία αυτά υπάρχουν πολλαπλά φαινόμενα απάτης ή διευκολύνονται σε αυτά τα σημεία τομής φαινόμενα απάτης. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι αυτή απάτηση, απλούστευση σε συνδυασμό με έναν αποκεντρωμένο σχεδιασμό δίνει ευρύ περιθώριο για διαφθορά και κατάχρηση. Είναι σημαντικό λοιπόν κύριε Επίτροπε τις ε, σχεδιαστείς μεταρρυθμίσεις να ε, λάβουμε υπόψη τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις γιατί ε, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούμε μελλοντικά με μία αύξηση των φαινομένων κατάχρησης. Ευχαριστούμε πολύ κύριε συνάδελφε. Ε, λυπούμε που δεν ήταν δυνατόν να μιλήσουν όλοι όσοι ήθελαν να πάρουν το λόγο στα πλαίσια διαδικασία Catch the Eye, αλλά έχουμε μια μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Επόμενος ε, ο εκ μέρους της Επιτροπής, ε, το λόγο έχει ο κύριος ε, Χάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πολύ πλατιά και πολύ στρατευμένη αυτή συζήτηση. Ο κ. Φεραίρα έχει φύγει ε, δυστυχώς από την αίθουσα. Ε, είπε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερες βάθος με το θέμα αυτό. Ωστόσο, όπως έχει υποθεί, η πόλη είναι η σημαντικότερη κληρονομιά του ανθρώπου. Και δεν μπορούμε να προσθέσουμε εδώ τίποτα παραπάνω γιατί πραγματικά τα αστικά κέντρα είναι τα δεδομένα εργαστήρια για τις κοινωνικές εξελίξεις, τις θετικές και τις αρνητικές. Ως εκ τούτου θα πρέπει η ανάπτυξη της Ευρώπης να στηριχθεί στην ανάπτυξη των αστικών κέντρων και πολλούς από τους στόχους του 2020 ε, μπορούν να επιτευχθούν μόνο εφόσον ασχοληθούμε με τα προβλήματα των πόλεων. Ο εδαφικό τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντικό ε, και πραγματικά είμαι ευγνώμων που αφιερώσετε μια ιδιαίτερη έκθεση εδώ. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη, ωστόσο ε, προσαρμοσμένες τους, στα, στις κανονιστικές μας δυνατότητες εργαλεία. Εδώ θα πρέπει να ισχύσει η αρχή της ε, διακυβέρνησης, η οποία προτείναμε ως Επιτροπή, η οποία πρόκειται να συνεχιστεί και στους, ε, στις κανονιστικές διατάξεις, στα regulations, και θα πρέπει να είναι καθοριστική, ε, και καθοριστικό εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας και το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επίσης έχει τύχει της προσοχής σας. Όταν ανέλαβα το αξίωμά μου, ε, χρειαζόταν να πείσουμε τις νέες χώρες μέλη για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα της ενέργειας. Εν τω μεταξύ έχει γίνει κοινή πεποίθηση πόσο μεγάλη είναι η αξία της ενεργειακής πολιτικής και ελπίζω στις ε, μελλοντικές ε, regulations να δοθεί επαρκής χρηματοδότηση για όλα αυτά τα θέματα. Τώρα, ε, εν συντομία στο Ταμείο Ελληνικής. Και εδώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας και όπως ε, ήδη εξήγηλα, σε ε, τις προσεχείς εβδομάδες θα υποβάλουμε μια σχετική πρόταση. Ωστόσο, θα πρέπει να σας απογοητεύσω ως προς το εξής. Δεν θα είναι δυνατό το Ταμείο Αλληλεγγύης ε, να ενταχθεί στο κανονικό προπολογισμό, αλλά θα συνεχίσει να εξυπηρετείται εκτός του προπολογισμού με τη βεβαίως ε, αναγκαία προηγούμενη διαδικασία της ε, αξιολόγησης όσον αφορά τις τάξεις μεγέθους χρημάτων κονδυλίων που είναι αναγκαίες. Ε, η πρόταση, υπάρχει πρόταση η αξιολόγηση των φυσικών καταστροφών να γίνει μελλοντικά πιο εύκολη. Ε, παρακαλώ ε, λίγο να χαμηλώσετε τα κινητά. Γιατί ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτρο που θα το θέμα αυτό για να μην χρειάζεται να το πω εγώ. Λοιπόν, ε, όσον αφορά το Ταμείο ε, θα υποβάλουμε μια πρόταση η οποία έχει σαν σκοπό η αξιολόγηση των φυσικών ε, καταστροφών να γίνεται πιο εύκολη ούτως ώστε στην πράξη η πιθανότητα να ικανοποιούνται τα αιτήματα να αυξάνεται. Θα υπάρξει λοιπόν μια απλούστευση και απλούστευση υπό την έννοια της ε, μεγαλύτερης εξασφάλισης των ε, πληγέντων όσον αφορά την καταβολή αποζημιώσεων. Γιατί αυτό το επιτάσσει η αρχή μιας ε, έντιμης, σωστής αντιμετώπισης των θυμάτων των φυσικών καταστροφών, ούτως να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Ε, τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της ε, πρόληψης, θεωρώ ότι και αυτή είναι μια σημαντική πτυχή στην οποία θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο μέλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τις διάφορες επισημάνσεις όσον αφορά τις πραγματεύσεις για το MFF. Ε, εδώ δεν θέλαμε να προσθέσουμε τίποτα. Η στάση της, η είναι ξεκάθαρη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για την επισήμανση της αναγκαίας επικέντρωση σε ορισμένα θέματα ε, καθώς και ε, στην ανάγκη μιας καλύτερης επικοινωνιακής πολιτικής. Γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό ε, να θεωρήσουμε ότι αυτή είναι μια πολιτική στην οποία θα πρέπει να, το να επενδύουμε στις υποδομές. Αυτή είναι μια έκφραση έμπρακτης αλληλεγγύης Ε, τα χρήματα αυτά θα πρέπει να πάνε στις φτωχότερες ε, περιοχές. Αλλά το πώς θα γίνονται οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να ενταχθεί σε μια, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επενδυτικής ε, πολιτικής. Ε, και εδώ θα πρέπει να καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες γιατί θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό σωστά διανεμημένα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής είναι σε θέση να εξασφαλίσουν θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλική σας επισήμανση ότι τα κινητά θα πρέπει να χαμηλώσουν. Ο κύριος Κοτσολίνο είναι ο επόμενος ομιλητής. Παρακαλώ. Εδώ αναπτύχθηκαν δύο ουσιώδεις ε, αρχές τις οποίες ανέπτυξαν και οι συνάδελφοι οι οποίοι και μίλησαν εδώ αλλά και αυτοί οι οποίοι ε, βοήθησαν στην προετοιμασία της έκθεσης. Πώς είναι δυνατόν ε, να αναπτύξουμε στο μέλλον της ε, πόλης είναι δεδομένο ότι τουλάχιστον 5% ε, των ε, πόρων του νέου προγραμματισμού των διαφορετικών ταμείων μπορεί να αφιερωθεί σε ένα πρόγραμμα ε, αναβάθμισης των πόλεων. Αυτό είναι ένα καινοτόμο στοιχείο το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, αναπτυχθεί περαιτέρω και από την ίδια τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής και της τάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά ε, θα πρέπει να κάνουμε και μία τρίτη σκέψη που είναι νομίζω πολύ ισχυρή και στη συζήτηση. Το θέμα της, ε, των πόλεων μας οδηγεί σε ένα άλλο γενικότερο θέμα. Είναι ε, σε θέση η Ευρώπη να μπει σε ένα δρόμο ανάπτυξης. Θα πρέπει να βρεθεί διέξοδος από το πρόβλημα το οποίο κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε ε, τα τον επόμενο χρόνο, τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερους πόρους στο νέο προπολογισμό, όπως κατεδείχθη σαφώς από τη συζήτηση. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε ε, ε, ε, μονάχα ασκήσεις επί χάρτου. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε τέτοιες ασκήσεις και τέτοιους πειραματισμούς όσον αφορά τα project bonds και τέτοιου είδους σκέψεις. Επίσης και βεβαίως εδώ αναγνωρίζω την ευαισθησία της Επιτροπής και του Επιτρόπου να δοθεί μία μια ισχυρότερη πολιτική βάση. Τούτη τη στιγμή δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη ε, να συμβάλλει αποφασιστικά στο θέμα αυτό χωρίς μια ικανή νομική βάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Επόμενο ομιλητή για δύο λεπτά ο κύριο Βόν. Παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος στις τελικές μου παρατηρήσει να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη συνεισφορά του να ευχαριστήσω επίσης και τους συναδέλφους για τις ιδέες τους, να ευχαριστήσω τους Κιώδης και την Επιτροπή Απασχόλησης, η οποία εξέδωσε τη δική της νομοδότηση. Υπάρχει τη στήριξη για την ιδέα να συνδυάσουμε τις πιστώσεις όπου αυτό είναι εφικτό. Πολλά μένει βέβαια να γίνουν ακόμα έτσι ώστε να συνδυαστούν και οι κανόνες με τους οποίους χορηγούνται οι πιστώσεις από διαφορετικά ταμεία, αν το πετύχουμε αυτό. Αυτό θα είναι θετικό για τους, ε, ε, αυτούς που ετούνται στήριξης. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους του 2020. Αυτοί οι οποίοι καταφέρνουν αιτήσει και θέλουν να απλοποιηθεί η διαδικασία είναι θα έλεγα αυτοί που θα κερδίσουν από την ευελιξία η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζει από εδώ και πέρα τις διαδικασίες. Νομίζω ότι και κάποιες από τις προτάσεις της εκθέσεώς μου για το συνδυασμό των ταμείων μπορούν να βοηθήσουν. Πολλές περιφέρειες εξετάζουν αυτούς τους μηχανισμούς συνδυασμού των πιστώσεων, αλλά και βέβαια κάποιες άλλες περιφέρειες έχουν μείνει σχετικά πίσω. Πάντως εκτός κοινού πλαισίου υπάρχουν και άλλα ταμεία όπως το Horizon 2020. Πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά, να συνεργαστούμε με τις τοπικές αρχές, να ανταλλάξουμε χρηστές πρακτικές και να επηρεάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν το κάνουμε αυτό, τότε οι περιφέρειες θα βοηθήσουν και θα βοηθηθούν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επόμενη ομιλήτρια για δύο λεπτά είναι η κυρία Κολάρσκα Μπαμπίνσκα. Πολλή συζήτηση έχει γίνει για τις ε, πόλεις ε, οι οποίες θα πρέπει να αποτελήσουν μοχλό ανάπτυξης ε, των περιφερειών. Αλλά αυτό όμως δεν ισχύει πάντα. Οι γεωργικές περιφέρειες δυσκολεύονται πάρα πολύ ε, να ελκύσουν ε, νέες ε, επενδύσεις. Στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής η ανάπτυξη εφιούς ενέργειας θα είναι κεφαλαιόδους σημασίας. Γνωρίζουμε ότι στην Βόρεια Σουηδία μια περιοχή αναπήχθηκε μονάχα λόγω της ανάπτυξης της ενέργειας. Ε, δεν πρέπει να λησμονούμε επίσης ότι ε, για τις ε, περιοχές οι οποίες βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία και εν πάση περιπτώσει όπου υπάρχουν νέες ευκαιρίες να τις αδράξουμε. Βεβαίως θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν και ενέργειες όπως το φυσικό, το φυσικό αέριο, το συστολιθικό ε, αέριο που είναι πολύ σημαντικά για την ε, ανάπτυξη. Θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να δράξουμε τις ευκαιρίες που ε, παρουσιάζονται. Βεβαίως τα προγράμματα θα πρέπει να είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των περιφερειών έτσι ώστε να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Ε, δεν μιλάμε μονάχα ε, για ε, δαπάνη χρημάτων, δεν μας ενδιαφέρει μονάχα να δοθούν κάποια χρήματα ή κάποιοι πόροι. Θα πρέπει να ξέρουμε για τι περιοχή μιλάμε, τι είδους όραμα έχει αυτή η περιφέρεια, προς τα που θέλει να οδεύσει, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα πάντα με αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία συνάδελφε. Επόμενη ομιλήτρια για δύο λεπτά η κυρία Στάρα Σφεραγκούτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Σε αυτό το τελευταίο γύρο παρεμβάσεων θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν εκ μέρους της Επιτροπής για να υλοποιηθεί αυτή, αυτές οι έκθεσεις, καθώς και τον Επίτροπο ο οποίος ε, φάνηκε πολύ δεκτικός για αυτό το αίτημα ούτως ώστε να υπάρξει μια απλούστευση στη διαδικασία αυτή και να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια στην ε, υποβολή αιτήσεων. Ιδιαίτερως όσον αφορά τον ορισμό του τι συνιστά μια περιφερειακή καταστροφή. Μιλήσαμε για ένα λογικό δίκτυ που θα, πρέπει να, ε, θα μπορούσε να είναι το ΑΕΠ, αλλά ε, επίσης ε, οι ζημιές ε, που προκαλούνται για παράδειγμα στο τοπίο ή στο περιβάλλον και που ζημιώνουν τις, ε, τη ζωή της περιφέρειας αυτές. Πιστεύω ότι αν στο, το 2014 μπορέσουμε να έχουμε αυτόν τον κανονισμό τον οποίο εκπονεί η υποτροπή, αυτό θα είναι ευεργετικό για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα για να εκπληρωθεί η αρχή της αλληλεγγύης έτσι λοιπόν ο κύριος Επίτροπος ε, θα έχει σίγουρα την υποστήριξη αυτού του σώματος. Ευχαριστούμε πολύ κυρία συνάδελφε. Η κοινή συζήτηση για τις τέσσερις εκθέσεις έχει ολοκληρωθεί. Η ψηφορία και τις εκθέσεις των κυρίων ε, Κοτσολίνο Βος και Στάρας ε, Φερακούτ θα γίνει αύριο στις 12 ενώ η ψηφορία για την έκθεση της κυρίας ε, Μπομπίνσκα θα γίνει την Τετάρτη στις 12. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημέρης της διάταξης. Ακολουθεί η έκθεση του κυρίου Μπερλινγκουέρ